Bien, puisque Λοιπόν, σα προτείνω να περάσουμε στο σημείο 5, διότι έχει φτάσει ο αρμόδιο εισηγητή, το σχέδιο στατηγικών επενδύσεων και το θέμα τη νομική βάση σε ό,τι αφορά την τροποποίηση των κανονισμών μας. Έχουμε κάνει ανταλλαγές απόψεων ήδη με την Επιτροπή, τον Πρόεδρο της Κομισιόν ο οποίος έδειξε άμεσο ενδιαφέρον για το, την πρόθεση του θέματος αυτού και είχαμε συμφωνήσει να συνεργαστούμε σε επίπεδο απόλυτης ισότητα με την Επιτροπή ΕΚΟΝ χρησιμοποιώντας το άρθρο 54 του κανονισμού χρησιμοποιώντας το σύστημα των συνεισηγητών που θα είναι ο κύριος Όλμπρεχτ από την δική μας πλευρά διακόπτει ο πρόεδρος Συγγνώμη. Θα είναι ο κύριος Φερνάντης, ο εισηγητής μας. Αποφασίστηκε χθε από εμάς. Πάνει καλός, λέει ο πρόεδρος, οπότε ο κύριος Φερνάντες θα είναι ο αρμόδιος για την Επιτροπή Προϋπολογισμών και ο κύριος Μπούλμαν για την Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων. Και υπάρχουν και επιτροπές οι οποίες συνδέονται βάσει του άρθρου 54, οι επιτροπές Ήτρε και Τραν και επίσης οι Επιτροπές Απασχόλησης και Ελέγχου του Προϋπολογισμού βάσει του άρθρου 53α θα έχουν πρόσβαση στον τριγωνικό διάλογο για τα άρθρα που τις εμπλέκουν. Αναφέρθηκε επίσης και η δημιουργία μιας ομάδας συντονισμού ώστε να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η συνεκτικότητα κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας και για να παρακολουθηθεί το θέμα αυτό του Ταμείου Επενδύσεων σε επίπεδο Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την συνεργασία των Επιτροπών. Η Συνέλευση των Πρόεδρων δεν έχει λάβει ακόμα αποφάσει. Ελπίζουμε ότι σήμερα θα πάρουμε το πράσινο φω για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. χθε. υπεγράφηκε μια επιστολή προς την Συνέλευση των Πρόεδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών η οποία θα, θα διαβιβαστεί στην σημερινή συνεδρίαση των Πρόεδρων των Πολιτικών Ομάδων. Και για να μην χρονοτριβήσουμε, ίσως θα χρειαστεί να κάνουμε μια έκτακτη συνεδρίαση την Δευτέρα 9 του μηνός, όχι 8, 9 του μηνός, στο Στρασβούργο. Εφόσον έχουμε τη σύμφωνη γνώμη της Οικονομικής Επιτροπής βέβαια. Κύριε Φερνάντσου. Έχετε να κάνετε κάποια σχόλια. σε σχέση με την ε, ανάληψη της εισηγεσίας από τη δική σας πλευρά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα πορτογαλικά. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας που για μένα είναι πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν τη δημιουργία της ε, απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την οικονομική ανάκαμψη θα πρέπει να υποστηρίξουν το σχέδιο Juncker. Υποθέτω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες υποστηρίζουν τους στόχους και την ιδέα του Ταμείου Επενδύσεων. Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα προσελκύσει και ιδιωτικού πόρους για να επιτύχουμε το στόχο της ανάκαμψη και της απασχόλησης. Είναι σφιχτό το χρονοδιάγραμμα, αυτό θα μας υποχρεώσει να εργαστούμε με έντονο τρόπο. Η ελπίδα μου είναι ότι στην Ολομέλεια του Ιουνίου θα μπορέσουμε να λάβουμε την τελική απόφαση μαζί με το Συμβούλιο σε επίπεδο πρώτης ανάγνωσης και αν ε, επιληθούν όλα τα προβλήματα αυτά στην πρώτη ανάγνωση και μπορούμε να έχουμε ήδη λειτουργικό αυτό το ε, εργαλείο ήδη τον Ιούνιο, αυτό θα είναι θετικό. Αλλά υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών εδώ θα έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και όπως είναι προφανές μαζί με την Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να λειτουργήσει σε επίπεδο απόλυτης ισότητος γιατί επελέγει ως ε, βάση το άρθρο 55 του κανονισμού μας. Η Επιτροπή μας παίζει σημαντικό ρόλο διότι πρόκειται για ένα ε, πρόγραμμα το οποίο προϋποθέτει προϋποθ, ε, τροποποίηση του προϋπολογισμού, διορθωτικό προϋπολογισμό και επίσης απαιτείται μια συνένεση που υποθέτω ότι υπάρχει ήδη σε σχέση με την υποστήριξη αυτής της καινοτόμας ιδέας η οποία θα έχει επιπτώσεις και στην εσωτερική αγορά. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν μια σειρά από ενέργειες και θα πρέπει εν τέλει να εξασφαλίσουμε ότι η λύση η οποία προτείνεται για τις γραμμές του προπολογισμού που θα χρησιμοποιηθούν ως εγγυήσεις για το Ταμείο αυτό, θα πρέπει να δούμε αν έχουμε κάποιες εναλλακτικές δυνατότητες για αυτές τις γραμμές του προϋπολογισμού. Κατανοούμε φυσικά ότι ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθούν κάποιες γραμμές από τον ορίζοντα 2020 και από τη διευκόλυνση Connecting Europe. Αλλά από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το σχέδιο επενδύσεων θα χρειαστούν περισσότεροι πόροι από αυτούς που έχουμε ήδη προβλέψει στις γραμμές αυτές του Connecting Europe και του Horizon 2020, το να αντιμετωπίσουμε και άλλες γραμμές του προϋπολογισμού για την παροχή εγγύησεων μπορεί να σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια τροποποίηση στον προϋπολογισμό. Μπορούν να προκύψουν λοιπόν και περαιτέρω προτάσεις τροποποίησης του προϋπολογισμού που θα ετύχαναν μεγαλύτερη συνέντευξη μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τέτοιε προτάσει είναι απόλυτα καλόδεκτες. Και φυσικά ο δικό μου ρόλο θα είναι να προσπαθήσω να επιζητήσω τη μέγιστη συνεργασία από την πλευρά των πολιτικών ομάδων ε, υπέρ ενό στόχου που όπω σα είπα προηγουμένω, πιστεύω ότι υποστηρίζεται από όλου επενδύσει, υπέρ τη οικονομικής ανάκαψης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρο. Η κυρία Γουάρδια Σαβάλ. Θέλετε να μας πείτε κάτι για τον διορθωτικό προϋπολογισμό υπαριθμών γιατί συνδέεται άμεσα με τη νομική αυτή βάση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Χωσέ και εγώ από ό,τι φαίνεται είμαστε προορισμένοι να δουλεύουμε μαζί, γιατί εγώ είμαι υπεύθυνη για την σοσιαλιστική ομάδα, οπότε έχω αναλάβει το πρόγραμμα επενδύσεων και επίσης το σχέδιο προϋπολογισμού παριθμονένα, οπότε για άλλη μια φορά είμαστε καταδικασμένοι να συνεργαστούμε. Πάντως ε, αυτό το οποίο παρουσιάζεται ως ε, πρόταση του Κοινοβουλίου λοιπόν για, για το πρώτο διορθωτικό του προπολογισμού ε, θα ακολουθήσει την συμφωνία η οποία θα κλειστεί όσον αφορά τον τρόπο χρηματοδότησης και όσον αφορά τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου όσον αφορά το Οπότε και εγώ θα πρέπει να σας τονίσω κάτι το οποίο το προείπε ο Μανουέλ. Μπορούμε να διατυπώσουμε μια εναλλακτική όσον αφορά την συμμετοχή στον προπολογισμό. Βεβαίω, ε, χρειάζεται πλειοψηφία εδώ και επίσης χρειάζεται μετά πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Οπότε ό,τι πρόταση γίνει για να αλλάξει το ε, δημοσιονομικό πλαίσιο ε, χρειάζεται την ομοφωνία στο Συμβούλιο. Οπότε και αυτοί που θεωρούν ότι αυτό το ταμείο μπορεί να ε, χρηματοδοτηθεί από την ε, εξωτερική πολιτική, από τη Γεωργία ή από αλλού, να το ξεχάσουν. Είμαστε στην κατηγορία 1α. Έχουμε πάρα πολλές ε, πιθανότητε εδώ, οπότε θα πρέπει να σκεφτούμε κάποια εναλλακτική άλλη που θα μπορούσε να είναι διαφορετικός τρόπος ανάπτυξη του Ταμείου τα επόμενα χρόνια. Και με το Euro Facility δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα για το 2015, ούτως ώστε να αλλάξουμε τις πιστώσεις υποχρεώσεων και επίσης δεν χρειάζεται να έχουμε τόσα χρήματα ως εγγύηση που είναι δεσμευμένη. Ε, πρόκειται για για κάποιο ρήτρα διαφύλαξη ε, που έχουμε αυτά τα δισεκατομμύρια εδώ. Οπότε αυτά και θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Είναι θυσίες τα οποία δεν συνδέονται ίσως άμεσα με τον προπολογισμό, αλλά είναι δική μας αρμοδιότητας και πιέζει ο χρόνος, μια που θα πρέπει να έχουμε έτοιμη την έκθεση περί τα τέλη του μηνό. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήταν σωστό Έχοντας αυτό το πρόγραμμα το οποίο αφορά την ε, απασχόληση και την ε, ανάπτυξη και να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τρία θεσμικά όργανα μπορούν να αποφασίσουν ε, άμεσα. Ακριβώς γιατί πιέζει το θέμα. Κύριε Γκρέσλε, κύριε Πρόεδρε, ο Αντιπρόεδρος Κατάινεν μας επισκέφθηκε στην Επιτροπή μας. Τα συζητήσαμε και στην Ολομέλεια και έχω να πω ότι τα είπαμε και τα είπαμε, αλλά απάντηση δεν δόθηκε. Οπότε θα πρέπει να καταρτήσουμε αυτό το ερωτηματικό, να έχει συγκεκριμένη προθεσμία η γραμματεία και να ελπίσουμε ότι θα υπάρξει κάποια απάντηση τουλάχιστον τότε. Γιατί πάρα πολύ δύσκολο να κατεβάσουμε το μυαλό μα ένα νομοθέτημα όταν έχουμε κάποια βασικά ερωτήματα τα οποία ακόμα εκκρεμούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια προ τον ε, εισηγητή για το έργο του. Ευχαριστώ, λέει ο Ξέρω, ξέρω πόσο πιέζουν τα πράγματα και γι' αυτό ακριβώς και εγώ θα ήθελα να έχουμε αυτή την ε, ε, έκτακτη συνεδρίαση το, τη, τη Δευτέρα το βράδυ στο Στασβούργο με του συναδέλφου της ΕΚΟΝ. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στην κυρία Τομά, η οποία έχει κάποια υποχρέωση και πρέπει να φύγει όπου να είναι. Για πετε μα, πώς λέτε τα θέματα όσον αφορά αυτή την ε, τροποποίηση του πολιτού δημοσιονομικό πλαισίο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμπαθάτε με γιατί πρέπει να φύγω και σας αλλάζω και σειρά στη μέση διάταξη. Τώρα όσον αφορά την ε, τροποποίηση αυτή, ε, συνεργάζεται μαζί μου ο κύριος ε, Όλμπριχτ, ο οποίος και εκείνος μπορεί να με συμπληρώσει και είχαμε μια υστέρηση, καθυστέρηση τέλο πάντων μετά από την αργοπορημένη ψηφορία του πολιτούς πλαισίου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και όσον αφορά τους πόρους αυτούς της συνδιαχείρισης, αφορούσαν τα λειτουργικά προγράμματα, ε, πρέπει να, τρέξουν, πρέπει να, να, να στις 31 Δωδεκάτου από την Επιτροπή, είπαμε, γιατί έχουμε 13% τα οποία έχουν μεταφερθεί, από το 14% στο 15% και 47% ε, δεν καλύπτονται. Δηλαδή από αυτό το πρόγραμμα αυτοί οι πόροι έπρεπε να έχουν εγκριθεί 31 δωδεκάτου, Αλλά τώρα θα πρέπει να μεταφερθούν ως ε, πιστώσεις υποχρεώσεων στην επόμενη χρήση. Οπότε έχουμε τώρα το άρθρο 19 του που μας επιτρέπει να κάνουμε αυτή την ενέργεια όσον αφορά το πολιετές πλαίσιο και να σας πω με παραδείγματα για να καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι το πρόγραμμα. Είναι 99% των ε, προγραμμάτων για την Τσεχία, ας πούμε, ε, θίγονται από την υπόθεση. 59 και κάτι της εκατό των προγραμμάτων που αφορούν την Βρετανία και 66 και 5% για την Ιταλία. Κάποια παραδείγματα είναι που να σας δείξουν πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Επομένως πρόκειται για αυτή την τροποποίηση και αναθεώρηση που τελικά πρέπει να γίνει για να μην χαθούν αυτοί οι πόροι και να μπορέσουν να εκταμιευθούν. Και Βλέπω ότι είναι τεχνικού χαρακτήρα αυτή η τροποποίηση, η αναθεώρηση του πολίτους πλασίου. Οπότε και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να βραδύνουμε. Γιατί έτσι θα μπερδευτούν τα πράγματα από πλευράς κοινοβουλίου. Θα πρέπει το σημαντικό δυνατόν να προχωρήσουμε. Οπότε να επιληθεί το πρόβλημα. Τώρα, να μην ξεχνούμε ότι με αυτή την πρόταση της αναθεώρησης του πολιτού πλαισίου αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα των πληρωμών, διότι ξαφνικά τώρα μας προκύπτει μια χρήση που έχει μεταφερθεί από τις πιστώσεις πληρωμών. Όμως τώρα θα γίνει κάποια σόρευση πάρα πολύ πιθανό και οπότε όλα μετά ρισκάρουμε να πάνε στο 17 ή στο Άρα θα πρέπει χωρίς καθυστέρηση να προχωρήσουμε για την ευκαιρία να τονίσουμε σε Κομισιόν και Συμβούλιο ότι ε, ε, από τη μία μεριά έχουμε αυτό το, το, θεματολόγιο το πάντων για την κρίση των πληρωμών και από την άλλη μεριά έχουμε αυτή την αναθεώρηση του πολιτούς πλαισίου. Οπότε σε σχέση με το που λέει το ΕΛΚ. Λένε να γίνει διάμεση αναθεώρηση, άλλοι λένε μετεκλογική αναθεώρηση. Τέλος πάντων, τώρα να μην το αναλύσουμε πάλι. Αλλά θα πρέπει να γίνει αυτή η αναθεώρηση, Πρόεδρε. Οπότε ήρθε η ώρα, ήρθε η ευκαιρία να οργανωθούμε στο Κοινοβούλιο και εδώ στην Επιτροπή μας όσον αφορά το πώς θα μεθοδεύσουμε αυτή την αναθεώρηση. Κύριε Όλμπριχτ. Πρόεδρε, να μην επαναλάβω όλα όσα ακούσαμε ήδη. Να πω ότι καταρχάς υπάρχουν τριών ειδών προγράμματα σε ό,τι αφορά το επίπεδο δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχάς, τα προγράμματα τα οποία έχουν αναλυθεί και έχουν γίνει αποδεικτά. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα από το 2014. Και υπάρχει ο κανόνας νησιν 3 ε, για τα προγράμματα αυτά. Τα προγράμματα που έχουν γίνει αποδεκτά δηλαδή είναι στο νησιν 3. Ε, μέχρι το 2017. Ύστερα τα προγράμματα τα οποία δεν έχουν γίνει αποδεκτά αλλά είναι έτοιμα. Αυτό που ονομάζουμε carry τα οποία θα μεταφερθούν αυτόματα στο επόμενο έτος, το 2015. Και φυσικά και εδώ γίνεται αποδεκτός ο κανονάς Νίσιν 3, αλλά με αρχή το 2015 έως το 2018. Και τρίτη κατηγορία προγραμμάτων, τα οποία δεν έχουν γίνει αποδεκτά το 2014. Και φυσικά υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν τα χρήματα. Πρόταση λοιπόν είναι να μεταφορθούν οι δεσμεύσει, όχι οι πληρωμέ, οι δεσμεύσει από το 2014 στο 2015 εκτός από τα προγράμματα που έχουν τον κανόνα νήσιν 2 για το πρόγραμμα για το άσυλο. το Ταμείο για το Άσυλο και το Ταμείο για την Εσωτερική Ασφάλεια. Υπάρχει πρόταση λοιπόν να μεταφερθεί στο 15, 16, 17. Να σας υπενθυμίσω ότι το πρόγραμμα αυτό έχει τον κανόνα νησιν 2, αλλά ποτέ δεν γίνεται αποδεκτό τον πρώτο, το πρώτο έτος. Αν μεταφερθεί λοιπόν το 2015, το νησιν 2 ξεκινάει το 2016. Από αυτά που ξεκινάνε το 2016, το νησιν 2 θα ξεκινήσει από την επόμενη χρονιά. Τα προγράμματα στο 1α μεταφέρεται από το 14 στο 15 με την εξαίρεση του εργαλείου διασυνοριακού και ευρωπαϊκής γειτονίας που πάει στο 2017. Αυτό είναι λοιπόν το πρόβλημα με τον ε, κανονισμό συντρία. Άρα, συνοψίζοντας, είναι τεχνικό το θέμα. Το ερώτημα που έθεσε ο συνεισηγητής είναι ποια είναι ο αντίκτυπος της πληρωμές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ενημερώνει ότι επισήμως δεν υπάρχει άμεση επιρροή για τις πληρωμές στην παρούσα φάση, αλλά οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να μπουν και αυτό είναι το πρώτο στοιχείο, και να συμπεριληφθούν για τον προπολογισμό 2016. Τεχνικό μεν, αλλά επηρεάζει και τον προπολογισμό του 2015 και του 2016 και του 2017 σε ό,τι αφορά μία περίπτωση το πρόγραμμα για το άσυλο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις ε, εξηγήσεις αυτές. 26 Φεβρουαρίου μπορείτε να καταθέσετε την τροπολογία σας και 11 Μαρτίου θα έχουμε την προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Και 1 Απριλίου θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες. Μιλήσατε και τον DAB 2. Το διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 2. Σας ακούω με μεγάλη προσοχή και αυτό σε σχέση με μια συζήτηση η οποία θα έχει ιδιαίτερα τεχνικό χαρακτήρα. Δεν πρέπει να χάσουμε από τα μάτια μας την ουσία. Ο στόχος μας είναι η ανάπτυξη και η απασχόληση. Μιλάμε και πάλι για πιστώσεις πληρωμών και δεν λέμε τίποτα για τους πόρους, για τα έσοδα. Θα πρέπει και αυτό το θέμα να το λύσουμε κάποια στιγμή. Παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να πείσουμε κάποια στιγμή το Συμβούλιο να, να εξασφαλίσουμε ότι θα τροφοδοτείτε ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Μα στην έκθεση που θα παρουσιάσουμε για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα το υποστήριξω αυτό. Όπω είπατε, να έρχονται τα πρόστιμα από τα κράτη-μέλη στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να πάρουμε χρήματα από το Connecting Europe και από την έρευνα αυτό μου δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Δεν είναι ο τρόπο με τον οποίο θα δημιουργήσουμε συνθήκε ανάπτυξη και απασχόληση. σω πρέπει να βρούμε αυτά τα χρήματα κάπου αλλού. Ο μηχανισμό συνεπέδεται 10 από, αυτούς τους, ε, από αυτέ τι θέσει του προπολογισμού και θα σα δώσω 150. Περνάμε στον διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 2. Κυρία Γουάρια Σαγάλ πάλι. Δεν έχω πολλά να πω για το ΔΑΒ 2, τον διορθωτικό το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 2. Πρόκειται για μεταφορά πιστώσεων από προγράμματα που δεν μπόρεσαν να εκτελεστούν το 2014 λόγω καθυστερήσεων στη χρηματοδότηση, στους ε, κανονισμούς των προγραμμάτων. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε αυτά τα 21 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρονται ως υποχρεώσεις στο 2015 και 2016 πώς θα καλυφθούν από πληρώσεις πληρωμών. Γιατί έμειναν χρήματα διαθέσιμα τα οποία δεν ε, εκταμιεύτηκαν για τα προγράμματα που έπρεπε και έτσι πληρώθηκαν προηγούμενα ε, χρέη. Αλλά ήδη το 2014 είχαμε φτάσει στα 25 δισεκατομμύρια οφειλόμενα ποσά. Το θέμα είναι πώς θα τροποποιηθεί αυτό πώς θα αντιμετωπιστεί στον προϋπολογισμό του 2015. Σήμερα λέγεται ότι θα βελτιωθεί η προχρηματοδότηση για την εγγύηση για τους νέους, αλλά κάθε φορά που υπάρχει μια νέα είδηση, όλα αυτά σημαίνει ότι θα επιδεινωθεί η κρίση των ραλ, των μη εκταμιευθέντων ποσών του 2015-2016. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν υπόψη μας το σχέδιο της Κομισιόν για να λυθεί το πρόβλημα των απλήρωτων ποσών και αν θέλουμε να διατηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας, να τις στηρίσουμε και το ελπίζω αυτό, θα πρέπει να κάνουμε και τροποποίηση στις πιστώσεις πληρωμών και να αυξήσουμε τις πιστώσεις πληρωμών για να καλυφθούν αυτά τα ποσά τα οποία οφείλονται ακόμα. Για τις πληρωμές χρειάζεται συνέπεια από τη δική μας πλευρά και θα πρέπει να πάρουμε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να πιέσουμε το Συμβούλιο να λάβει υπόψη την ανάγκη ότι πρέπει να πληρωθούν οι οφειλόμενοι λογαριασμοί. Γιατί το Σύριο κερβασίζεται βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Θα πρέπει να μπορούμε να κινητοποιήσουμε τις εγγύησεις, εάν αυτό είναι απαραίτητο, αλλά πρέπει οι ιδιώτες επενδυτές για να συμβάλλουν σε αυτό το εγχείρημα πρέπει να έχουν πράγματι την βεβαίωση ότι εάν χρειαστεί οι εγγύησεις αυτές θα πρέπει να υπάρχουν για να κινητοποιηθούν. Σήμερα η Κομισιόν είναι... Θα πρέπει η Κομισιόν να το αποδείξει αυτό με το να πληρώνει με αρζάν κοντά, με ρευστό χρήμα της υποχρέωσης Ο κύριος Μόντι θα έρθει σε λίγα λεπτά. Έχει έρθει βέβαια ο κύριος Λαμασούρ. για την έκθεση Γουάρδια Σαβάλ και τα σχόλια που μας ανέφερε και σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Τωμάκη και ο κύριος θα έχετε κάποια σχόλια θα πρέπει να είναι σύντομη αυτή η ανταλλαγή απόψε γιατί έρχεται ο Σολούπο ο κύριος Μόντι κανείς δεν θέλει το λόγο όμως Oui, on va... On va suspendre quelques instants. Θα διακόψουμε τη συνεδρίαση. Relatif au fonds d'ajustement à la globalisation. Donc, je suspends la séance. Διακόπτω λιγάκι τη συνεδρίαση μέχρι την έλευση του κυρίου Μόντι. Mes chers collègues, je vous invite à regagner votre place. Καθίστε και πάλι αγαπητοί συνάδελφοι, αν θέλετε. La séance est reprise. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών έχει τη μεγάλη τιμή να υποδεχθεί τον καθηγητή Μάριο Μόντι, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία της πρώτης ενδιάμεσης εκθέσεως τα οποία έχουν παρουσιαστεί ήδη και στη συνέλευση των Πρόεδρων. Πρόκειται για τις εργασίες οι οποίες έχουν γίνει στα πλαίσια της ομάδας υψηλού επίπεδου για τους ίδιους πόρους και που προσπαθεί με τον τρόπο αυτό να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους ίδιους πόρους. Σήμερα έχει έλθει μαζί με τρεις εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Αλάν Μασούρ, τον οποίο χαιρετίζω, τον Ιβο Καλτσίν, τον οποίο επίσης χαιρετίζω, και τον Γκί Φερχοφ Στάτ, ο οποίος όμως είναι σε κάποιο βρυξελιώτικο μποτιλιάρισμα και θα έρθει μάλλον γύρω στις 10. Θα ήθελα να υπογραμμίσω την πολιτική σημασία των εργασιών αυτής της ομάδος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί όταν μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει μία αύξηση των ε, πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα μπορέσει να επιβάλλει ευρωπαϊκή φορολογία θα αλλάξει εκ το σχήμα της, ευρωπαϊκής, της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να συζητάμε μονάχα για τα θέματα των δαπανών, να κάνουμε συνδιαλλαγές και τριγωνικούς διαλόγους με το Συμβούλιο, όχι για τις υποχρεώσεις που συνάπτονται, αλλά μόνο για τις πληρωμές και ουσιαστικά για τις ισορρευόμενες καθυστερήσεις πληρωμών. Αυτό είναι ένα εγχείρημα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό για μας και φυσικά δεν λύνει τα ουσιαστικά προβλήματα ανταγωνιστικότητος ανάπτυξης και απασχόλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, εμείς αποδίδουμε τη μεγαλύτερη δυνατή σημασία στο έργο της ομάδος σας, κύριε Μόντι, και σας δίνω στο λόγο. Περιμένουμε με μεγάλη αδημονία την ε, ομιλία σας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών, είναι μια στιγμή μεγάλης σημασίας για τη δραστηριότητα της ομάδος της οποίας ηγούμε και για μένα τον ίδιο. Είναι πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή που έρχομαι ενώπιον της Επιτροπής σα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Προϋπολογισμών ιδίω έχουν αποκτήσει ένα ιδιαίτερο ρόλο, ένα εξόχως σημαντικό ρόλο σε όλη τη συζήτηση για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν, βρισκόμαστε τώρα στην καρδιά της ατμομηχανής για την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά αυτό συμπεριλαμβάνει τα πιο σημαντικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την χρηματοδότηση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει, υπέχει δουλείες ως προς τις άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα για την ευκαιρία αυτή να ανταλλάξω απόψεις μαζί σας. Μετά από τις πολύ εξαιρετικές διαπραγματεύσεις για τον ετήσιο προϋπολογισμό 2014-2015 και μετά την συμφωνία της τελευταίας στιγμής του Δεκέμβριο, είναι καλή η περίσταση να κοιτάξουμε τα πιο διορθωτικά και μακροπρόθεσμα στοιχεία που μας αποτελούν πρόκληση για τον προϋπολογισμό. Όπως θα ξέρετε, ήδη είχα την ευκαιρία να συζητήσω με την διάσκεψη των Προέδρων τις αρχές του Ιανουαρίου και να παρουσιάσω την πρώτη αξιολόγηση της ε, ομάδας υψηλού επίπεδου για τις ίδιους πόρους, η οποία και έγινε καλά αποδεκτή. Ελπίζω δε η σημερινή μας συζήτηση να επιτρέψει να προχωρήσουμε περαιτέρω. Ως μέλη της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού είστε οι βασικοί παράγοντες για τη συζήτηση για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Έχετε υποστηρίξει με συνέπειες ε, τις ε, μεταρρυθμίσεις, σημαντικές μεταρρυθμίσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ιδίων Πόρων. Είναι λοιπόν κρίσιμη σημασία. Πιστεύω να είσαστε ενήμεροι και να συμμετέχετε σε κάθε φάση των εργασιών της ομάδας. Ξέρουμε ποιε είναι οι δυσκολίε ε, οποιαδήποτε μεταρρύθμιση που προαπαιτεί ομοφωνία των κρατών μελών και μόνο αν το θέμα αυτό διατηρηθεί στην κορυφή της πολιτικής ατζέντα, θα καταφέρουμε να επιφέρουμε πραγματικές αλλαγές. Ως εκ τούτου, ελπίζω η πρώτη αξιολόγηση να έχει την προσοχή σας. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ως ένα εργαλείο για συζήτηση, ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω και ως σημείο αναφοράς για τις συζητήσεις σας. Να επαναλάβω λοιπόν στη συνέχεια τις βασικά περιστατικά το 2014 και να συνοψίσω τα βασικά μηνύματα της πρώτης αξιολόγησης, της πρώτης εκτίμησης. Και επί της βάσης αυτές μπορούμε να συζητήσουμε τις ε, θέσεις μας και το πώς θα προχωρήσουμε. Και με πολύ ανυπομονησία θέλω να ακούσω και τις δικές σας προτάσεις. Η ομάδα, όπως ξέρετε ξεκίνησε τις εργασίες της την άνοιξη του 2014 όταν το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχαν ορίσει τρία μέλη και είχαν από κοινού διορίσει τον πρόεδρο της ομάδας. Κάνοντας μου την τιμή να είμαι υποψήφιος. Η ομάδα λοιπόν ε, εκτέλεσε τα καθήκοντά της με καλή πίστη, με δέσμευση, με συνέχεια, παρά τις θεσμικές αλλαγές οι οποίες έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του 2014. Το Δεκέμβρη του 2014, μετά την ανάληψη των καθηκόντων της Επιτροπής Juncker, η ομάδα συναντήθηκε με τη νέα της σύνθεσης και συμφώνησε για την πρώτη της δημοσίευση παρά αυτά οι συζητήσει ήταν επικοδομητικέ, υπήρχε κλίμα συναδελφικότητα. Οι θέσει μας όμως δεν είναι ομογενεί απόλυτα. Τα μέλη, οι εμπειρίε του, οι τοποθέτηση του αντικατοπτρίζουν και την ποικιλία των συμφερόντων των ε, φορέων στα πλαίσια του προϋπολογισμού και όλοι ξέρετε πόσο μεγάλη είναι η πολυμορφία στο κλάδο αυτό. Αυτή η επικοδομητική λοιπόν πολυμορφία είναι απαραίτητη. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα αποκλεινόμενα συμφέροντα. Θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε για να υπάρξουν ε, χρήσιμες συστάσεις. Η ομάδα υψηλού επίπεδου λοιπόν έκανε την πρώτη της έκθεση αξιολόγησης πριν τα τέλη του 2014 και όπως προβλέπεται στην ε, κοινή δήλωση ίδιων πόρων του Νοεμβρίου 2013. Το πιστοποιητικό γέννησης, αν θέλετε, της ε, ομάδας. Η έκθεση, λοιπόν, κατατέθηκε παράλληλα στους προέδρους του Κοινοβουλίου, της Συμβουλίου και της Επιτροπής στις 17 Νοεμβρίου και επίσης την ίδια ημερομηνία δημοσιεύθηκε στο διαδικτύο. Στην έκθεση θεωρούμε ότι καταφέραμε να βρούμε μία ισορροπία στην πρώτη μας αξιολόγηση. Μία ισορροπία η οποία έπρεπε να παράγει τελικά ένα ισχυρό έγγραφο σε ό,τι αφορά την ανάλυση του υφιστάμενου συστήματος, αλλά παράλληλα να αποτελεί και μία ειλικρινή προσέγγιση σε ό,τι αφορά την αποφυγή προτάσεων για αλλαγή του τρέχοντος συστήματος. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι ήταν πολύ καλύτερο να αποστασιοποιηθούμε. Αυτή ήταν άλλωστε και εντολή που είχαμε λάβει. Να αποστασιοποιηθεί το κομμάτι της ανάλυσης, της διάγνωσης για τα θέματα του υφιστάμενου συστήματος από το επόμενο στάδιο. Τον εντοπισμό λύσεων, προτάσεων προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. όπως και οι συνάδελφοι, όπως ξέρουν καλά οι συνάδελφοι και της πρώτης ομάδας και της ταποποιημένης σύνθεσης της ομάδας, ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί για να μην παραβιάσουμε αυτή την ε, αρχή που διέπει τις εργασίες μας. Επειδή, κύριε Πρόεδρε, υπήρχαμε, υπήρχαν και στο κεφάλι μας ε, ήδη κάποιες σαφείς ιδέες για το πώς να αλλάξουμε το σύστημα. αν είχαμε ήδη εκφράσει τέτοιες ε, ιδέες, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ιδέες αυτές, αλλά αν τις είχαμε εκφράσει, το έγγραφο θα ήταν πιο ενδιαφέρον, λιγότερο άχρωμο αν θέλετε. Αλλά, αλλά, θα είχε προκαλέσει μία παραπλάνηση αν θέλετε γιατί κάποιος που βλέπει ποιε είναι αδυναμίε του υφιστάμενου κειμένου, αλλά ενδεχομένω να μην του άρεσαν οι συγκεκριμένες ιδέες, οι συγκεκριμένες προτάσεις που θα είχαν ε, συμπεριληφθεί, αυτό το άτομο λοιπόν, αυτό το θεσμικό όργανο, ενδεχομένως να είχε αποστασιοποιηθεί και από την αναλυτική περιγραφή των αδυναμιών του συστήματος. Πολύ απλά γιατί δεν θα του άρεσαν οι προτάσεις. Θέλαμε λοιπόν αμερόληπτη εξέταση να συμπεριληφθεί, αμερόληπτη αξιολόγηση του τρέχοντος συστήματος από όλους τους φορείς, χωρίς να μπλεχτούμε στις ιδέες και στις προτάσεις για το μέλλον. Θα υπογραμμίσω ένα κομμάτι όμως ότι σε αυτό το θεσμικό όργανο, σε αυτή την επιτροπή τη δική σα. η αξιολόγηση του τρέχοντος συστήματος, που δεν είναι και πολύ ευνοϊκή, δεν ξέρω αν το προσέξατε, είναι ομόφωνη αξιολόγηση. Άρα όλα τα μέλη της ομάδας, χωρίς εξαίρεση μετά από εξαρτητικές συζητήσεις, προσυπογράφουν την αξιολόγηση αυτή, την εκτίμηση αυτή. Και αυτό συμπεριλαμβάνει παρεπιπτόντως και τα τρία μέλη της ομάδας, τα οποία ορίστηκαν, διορίστηκαν από το Συμβούλιο. Είναι προκθαρτικό το έγγραφο. Γκρίζο και άχρωμο, σύμφωνοι. Αλλά η πολιτική σημασία του ότι εγκρίθηκε ομόφωνα πιστεύω ότι μας πάει ένα βήμα παραπάνω από ό,τι στο παρελθόν. Αποφύγαμε να είμαστε προκλητικοί, μεροληπτικοί, γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι χρειαζόμαστε να συμμετάσχουν όλοι οι φορείς, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, αν θέλουμε να αναθεωρήσουμε το σύστημα ίδιων πόρων. Όπως θα θυμάστε, είναι ένας τομέας όπου η νομοθεσία αποφασίζεται ομόφωνα. Αυτό προβλέπει επικύρωση σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές και ε, προαπαιτεί και έγκριση από το Κοινοβούλιο για τον εφαρμοστικό κανονισμό. Ήμασταν όμως πάρα πολύ σαφείς, ελπίζουμε τουλάχιστον, για το ποια είναι τα προβλήματα του τρέχοντος συστήματος και αφιερώσαμε ένα ιδιαίτερο τμήμα της ανάλυσης στις αδυναμίες του συστήματος. Τώρα, εν συντομία, να σας ε, παρουσιάσω το περιεχόμενο της πρώτης έκθεσης αξιολόγησης. Αυτή η έκθεση αποτελεί τη βάση για το έργο μας για το 2015-2016. Περιγράφει στην αρχή το τρέχον ε, χρηματοδοτικό σύστημα του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού που βασίζεται ε, στο σύστημα πιο πολύ εθνικών συνεισφορών παρά ιδίων πόρων. Περίπου 80% λοιπόν των εισόδων του προπολογισμού προέρχεται από άμεσες ε, συνεισφορές από τους εθνικούς ε, προϋπολογισμούς, 83% συγκεκριμένα το 2013. Είτε υπομορφή εθνικών συνεισφορών που υπολογίζονται βάσει του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, είτε υπομορφή ποσοστού της ε, βάσης ε, ΦΠΑ. Αυτό δεν ήταν πάντα έτσι. Έχει αλλάξει η σύνθεση των ιδίων πόρων πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και αυτό έχει κάνει τις ε, δημοσιονομικές διαπραγματεύσεις μεταξύ κρατών μελών ακόμα πιο έντονες και εστιαζόμαστε πιο πολύ στο αρκετά επιφανειακό στοιχείο των καθαρών ε, ισολογισμών. Πριν από δύο χρόνια είχα την ευκαιρία ως μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τότε είχα την ευκαιρία να δω εκ των έσω ποια είναι η φύση των διαπραγματεύσεων αυτών και να σας πω ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση η πιο ευγενής στιγμή της πολιτικής στη ζωή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Πιστεύω ότι η αντίληψη των πολιτών για το τι κάνει αυτή η περίεργη Ευρωπαϊκή Ένωση σε καμία περίπτωση δεν ε, εξοραίζεται με τη διαδικασία αυτή της διαπραγμάτευσης. Ε, σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις λοιπόν αυτές. Η έκθεση επίσης ε, υπενθυμίζει τις πρόσφατες προσπάθειες μεταρρυθμίσεις και υπενθυμίζει ότι οι δύο τελευταίες απόπειρες που έγιναν ε, κατά τις διαπραγματεύσεις του 2013-2014 2020 δεν κατάφεραν να μεταρρυθμίσουν την ουσία των προγραμμάτων και ουσιαστικά επέφεραν ίσον σημασία σε αλλαγές. Προκειμένου λοιπόν να προετοιμαστούμε για τα σημαντικά καθήκοντα του μέλλοντος, η έκθεση κοιτάει τα κριτήρια για ένα στεναρό σύστημα ίδιων πόρων και ευρύτερα θέματα πλαισίου, τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω προκειμένου να υπάρξουν οι συνθήκες για τη μεταρρύθμιση. Μεταξύ των κριτηρίων λοιπόν αυτών, που θα πρέπει να πληρούνται για να υπάρχει ένα εύρυθμο σύστημα ίδιων πόρων, θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή της δικαιοσύνης. Γιατί προφανώς αυτό περιλαμβάνει πάρα πολλούς, ε, πάρα πολλούς παράγοντες σε ό,τι αφορά θέματα διανομής και προκειμένου να υπάρχει και δημοσιονομική ισορροπία. Έχει πολιτικά φυσικά ιδιαίτερη σημασία και επηρεάζει τις ε, αντιλήψεις που επηρεάζουν τις πολιτικές αποφάσεις. Εν συντομία, αυτή η πρώτη έκθεση αναγνωρίζει τα μεγάλα εμπόδια για τη μεταρρύθμιση του τρέχοντος συστήματος. Αυτό δεν θα σας προκαλέσει ασφαλώς έκπληξη, αλλά επίσης αναζητά πρακτικές λύσεις βάσει διάφορων κριτηριών που θα πρέπει να βοηθήσουν στη λήψη μελλοντικών αποφάσεων βάση μιας ευρύτατης συζήτησης που θα περιλαμβάνει οικονομικά, θεσμικά, χρηματοοικονομικά και πολιτικά ζητήματα. Το συμπέρασμα λοιπόν το οποίο βγάζουμε στην παρούσα φάση προσωρινός είναι ότι δεν αρκεί να κοιτάξουμε τους διάφορους πόρους από τεχνική σκοπιά χωρίς να λάβουμε υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο. Επίσης, θα πρέπει να εξετάσουμε τις δυνάμεις που συντρέχουν και εξηγούν ποια θα είναι ενδεχομένως, η έκβαση μιας μεταρρύθμισης, αποτυχία ή επιτυχία. Άρα, πρέπει να κοιτάξουμε την πολιτική, τις πολιτικές σχέσεις και την πολιτική πορεία μιας τέτοια εξέλιξης. Μπορεί να έχετε σημειώσει τα διάφορα ερωτήματα τα οποία έχουμε θέσει και έχουμε διατυπώσει στην αξιολόγηση. Η εξέφραση απαντήσεων θα πρέπει να αποτελέσει κοινή προσπάθεια. Ιδιαιτέρως ε, επειδή κάποια από αυτά τα ζητήματα εμπίπτουν σε θεσμικά, θεσμικές αρμοδιότητες. Κύριε Πρόεδρε, θα κλείσω σε ό,τι στα θέματα διαθεσμικής συνεργασίας στο μέλλον. Η απόφαση να δημιουργηθεί η ομάδα αυτή υψηλού επίπεδου θα θυμάστε ότι ελήφθησε στις τελευταίες φάσεις της διαπραγμάτευσης για την προπολογισμό 2014-2020. Χάρη στην συνεχή υποστήριξή σας, προκειμένου να δοθεί η νέα πνοή στη συζήτηση για την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. και βλέπω ότι η ομάδα της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω αποτελεί λοιπόν πιο α, ζωντανή εκδοχή από την ταφή του σχεδίου. Και δεν τα λέω αυτά σε πνεύμα νεκροφιλίας, αλλά με μία συγκρατημένη αισιοδοξία, αν θέλετε. Ο παραδοσιακός τελικός προορισμός πολύ τολμηρών προτάσεων στην κοινωτική ιστορία, όπως ξέρουμε, το καλάθι των αχρήστων. Ήταν ε, λοιπόν εξαιρετική θεωρώ η ιδέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ιδιαιτέρως και κάποιων ε, εξεχουσών προσωπικότητων στο Κοινοβούλιο. Ήταν εξαιρετική λοιπόν η ιδέα που μας ε, ανάγκασε γιατί ήμουν και εγώ ακόμη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκείνη την εποχή να σοβαρευτούμε λίγο στην συμπροκειμένη περίπτωση και να ξεκινήσουμε μια διαδικασία γιατί δεν είναι τόσο σημαντικό να υπάρχει απλά μια ομάδα Πολλές φορές ε, συστήνονται ομάδες για να θάψουν πιο πολύ ένα ζήτημα παρά να το διαλευκάνουν. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ ότι το ένστικτο που επικράτησε ήταν πάρα πολύ ωφέλιμο και ήταν πραγματικά πολύ σκόπιμο. Το ότι δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα για τους ίδιους πόρους αντί να θαυτεί για άλλα 7 τουλάχιστον χρόνια το θέμα αυτό. Άρα, Συγχαρητήρια απευθύνω στους ε, δημιουργούς ε, της ε, ιδέας αυτής, στις διαπραγματεύσεις, παρά το γεγονός ότι αποτελούν ένα θύμα πλέον αυτής της εξαίρετης ιδέας. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι οι διαπραγματευτές ήταν ε, ενήμεροι και είχαν υπόψη τους ότι ο κλάδος των ε, εσόδων του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού ήταν ένα άλυτο ακόμα ζήτημα και αποφάσισαν λοιπόν να αντιμετωπίσουν κάποια από τα δημοσιονομικά ζητήματα προκειμένου να ξεκλειδώσουν κάποια από το δυναμικό του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Οι πιο πολλοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τολμώ να πω, συμφωνούν με την αντίληψη αυτή ότι ο ευρωπαϊκός προπολογισμός για την υποστήριξη των κοινών πολιτικών παραμένει ένας κλάδος που δεν χρησιμοποιεί το πλήρες δυναμικό του. Με μεγάλο ενδιαφέρον θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας απόψεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτό σε ό,τι αφορά μεταρρυθμίσεις από την πλευρά των ίδιων εσόδων. Θα θυμάστε ότι η κοινή διακήρυξη καλεί να διοργανωθεί διαθεσμική διάσκεψη με τα εθνικά κοινοβούλια. Ήταν πραγματικά μακρόπνοη αυτή η ιδέα. Τα εθνικά κοινοβούλια, τουλάχιστον θεωρητικά, είναι αυτά που είναι κατεξοχήν αρμόδια για τις προτάσεις, για τους ιδίους πόρους. Σε κάποιες περιπτώσεις, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ψυχολογικά, θεωρούν λοιπόν ότι είναι αρμόδια, αλλά στη πραγματικότητα τα εθνικά κοινοβούλια σπάνια έχουν την ευκαιρία να τα συζητήσουν αυτά σε βάθος. Είναι συχνά η επικύρωση τεχνικό ζήτημα και ουσιαστικά δεν οδηγεί σε ουσιαστική αλλαγή. Άρα η διάσκεψη το 2016 μεταξύ του Κοινοβουλίου του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων θα πρέπει να αποτελέσει μια ευκαιρία για πραγματική συζήτηση. Μια συζήτηση που δεν θα είναι εύκολη για κανέναν εμπλεκόμενο, αλλά που θα δώσει πραγματικά δημοκρατικές ε, ευκαιρίες. Είναι σημαντική η χρονική συγκυρία. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να λάβει χώρα πριν τη δημοσίευση της τελικής έκθεσης και των τελικών συστάσεων της ομάδας μας. Τα εθνικά κοινοβούλια δεν θα πρέπει απλά να σημειώσουν ποιες είναι οι συστάσεις της ομάδας ε, ίδιων πόρων που θα δημιουργηθεί μεταξύ των θεσμικών οργάνων, αλλά θα πρέπει να συμμετάσχουν άμεσα στην διαδικασία αυτή. Πιστεύω λοιπόν ότι η διάσκεψη αυτή θα πρέπει να λάβει χώρα όταν θα υπάρχει μια σαφής σχετικά προκαταρτική εικόνα του πού οδεύουμε και πού θέλουμε να οδεύσουμε για τις σημαντικές αυτές αλλαγές. Και να ακούσουμε και τις προτάσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων. Η ομάδα λοιπόν θα διοργανώσουν τις εργασίες της προκειμένου να είμαστε καλά προετοιμασμένοι για αυτή την διακοινωνική διάσκεψη παρά το γεγονός φυσικά ότι εσείς θα είσαστε οι πρωταγωνιστές αλλά θα είμαστε και ανοιχτοί για αλλαγές, γιατί το Κοινοβούλιο προφανώς έχει πολύ μεγάλη εμπειρία με διακοινοβουλευτικές διασκέψεις και είδα ότι ήταν θερμή η υποστήριξη της διάσκεψης των Προέδρων το Γενάρη για την διοργάνωση της διάσκεψης. Και τέλος, επιτρέψτε μου με ένα πολύ εγκάρδιο τρόπο, κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω ιδιαίτερος τα μέλη της ομάδας της οποίας προεδρεύω, τα οποία και διορίστηκαν τους κόλπους της ομάδας μας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Λαμασούρ, Φερχόφστατ, Καλφίν. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων που αποφασίστηκε εδώ στο Κοινοβούλιο παρά τις εξελίξεις ε, των θέσεων των προσωπικότητων αυτών τους επιτράπηκε να συνεισφέρουν και να συμβάλλουν σημαντικά στην εργασία μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Λέει ο Πρόεδρος. Merci pour euh, cette communication d'un rapport σας ευχαριστούμε για αυτή την ανακοίνωση όσον αφορά αυτή την προκαταρκτική έκθεση και καταλαβαίνουμε το ότι πρέπει να προχωρήσετε με μεγάλη προσοχή γιατί σίγουρα και πρόκειται για μια πάρα πολύ κρίσιμη πρόκληση. Οπότε και πρόκειται για μια βασικά κοινοβουλευτική πρωτοβουλία. Και τη μέρα που θα εμείς θα εγκρίνουμε την πρόταση αυτή, τότε τα εθνικά κοινοβούλια θα, θα σπεύσουν να εφαρμόσουν αυτό το οποίο προτείνατε, το οποίο θα είναι βέβαια για τους φορολογούμενους πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε που μας είπατε πώς προχωρήσατε, είμαστε στο πλάι σας. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Λαμαζούρα αν θέλει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίω, και 100% συμφωνούμε με την ε, άρτια ανάλυση του Πρόεδρου Μόντι. μεγάλη μας χαρά είδαμε ότι δέχθηκε αυτή την ε, ε, ευθύνη για αυτό το έργο που είναι πολύ δύσκολο. Πρόκειται για ένα θέμα που από πολιτικής πλευράς είναι σχεδόν αδύνατο να το διεξέλθει κανείς. Όμως πρέπει να πετύχουμε στο στόχο μας. Αδύνατον αλλά αναγκή. Επομένω θα τα καταφέρουμε. Και η Επιτροπή των Προϋπολογισμών γνωρίζει πόσο τούτο είναι αναγκαίο. Γιατί η κοινή γνώμη και δυστυχώς οι περισσότερες κυβερνήσεις δεν έχουν επίγνωση ότι σήμερα καμία νέα πολιτική, καμία νέα πρωτοβουλία δεν μπορεί να αποδώσει. Γιατί ξεκινούμε με 25 δις για κάποιες ε, οφειλές από τις προηγούμενες χρήσεις. Και οπότε, εάν δεν μπορέσουμε τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα να βρούμε μια λύση στο πρόβλημα της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών πολιτικών, ε, τότε αυτό θα είναι ο αργός θάνατος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο γίνεται σήμερα με την Ελλάδα και τις αγορές θα είναι απείρως χειρότερο για όλη την Ευρώπη εάν έχουμε αυτόν τον ε, αργό θάνατο. Ένα δεύτερο θέμα που θέλω να σας επισημάνω γιατί το ανέφερε ο Μαριμόντι αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό τα μέλη της Επιτροπής να το γνωρίζουν ότι από την πρώτη μέρα αυτό το θέμα το ανέλαβε το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή των Προπολογισμών. Και όταν λέω την αρχή, ενώ από το 2006. Όμως η Ευρωπαϊκή Οικοδόμηση απαιτεί μία ιόβιο υπομονή. Και τότε είχαμε τον κύριο Λεβαντόφσκι, ο οποίος προείδρευε της Επιτροπής των Προϋπολογισμών κατόπιν ήταν ο Ράινερ Μπέγκε που θα έρθει. Εγώ ήμουν εισηγητής και ο κύριος ε, Λεβαντόφσκι πήγε στην Επιτροπή μετά και ήταν εκείνος που στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, το έθεσε ότι χρειάζεται. Δηλαδή αυτή η μεταρρύθμιση που θα πρέπει να είναι μια πρώτη βάση για τις ε, εργασίες μας. Πολύ σημαντικό αυτό να το ξέρουμε. Και επίσης θα πρέπει να γνωρίζει η Επιτροπή των ότι η διάγνωση που έγινε από μας και κατευθυντήριες για αναζήτηση λύσεων που είχαμε προτείνει σε διάφορα ψηφίσματα ενσωματώθηκαν σε αυτήν την πρώτη αξιολόγηση που καταγράφει το τι έχει συμβεί. Κύριε Οπότε τελικά και τα άλλα θεσμικά όργανα και το Συμβούλιο παραδέχτηκαν αυτό το οποίο εμείς διαγνώσαμε ως ε, πρόβλημα στο σύστημα το οποίο δεν έχει διαφάνεια, είναι αντιδημοκρατικό και κανένα κοινοβούλιο δεν κάνει τέτοιου είδους ε, συζήτηση για τον προπολογισμό. Είναι αντιευρωπαϊκό αυτό το σύστημα. Είναι σαν να έχουμε στο Συμβούλιο 28 Θάτσερ. Αναποτελεσματικό θα είναι στο μέλλον μια που δεν υπάρχουν τα χρήματα. Και αυτό το οποίο επισημαίνεται σε αυτή την πρώτη αξιολόγηση αναφέρεται και ότι το σύστημα αυτό είναι άδικο. Γιατί όσο πιο ε, πλούσια είναι μια χώρα, τόσο λιγότερο συμβάλλει. Και οι λιγότερο πλούσιοι συμμετέχουν περισσότερο. Και αυτό όμως δεν το ξέρει κανείς. Ούτε στα εθνικά κοινοβούλια. Άγνοια. Δεν το ξέρουν οι Υπουργοί Οικονομικών και Προϋπολογισμών. Γιατί συνήθως είναι πρόκειται για ε, κάποιους τεχνοκράτες ε, της κυβέρνησης οι οποίοι κάνουν τις ε, διαπραγματεύσεις. Οπότε και εμείς κατεβάσαμε αυτές τις προτάσεις για τεχνητήριες γραμμές, λογικές, και ήρθαμε σε επαφή με τα Εθνικά Κοινοβούλια, κάτι το οποίο θα ξαναγίνει τώρα, ακριβώ όπω προτείνεται που πρότεινε ο κύριος Πρόντι, ο κύριος Μόντης. Και είπαμε ότι θα έχουμε τεχνητές γραμμέ αυτές για ένα σύστημα που θα είναι απλό, θα είναι δίκαιο. Δίκαιο και μεταξύ κρατών μελών και όσων αφορά του πολίτες, θα διακρίνεται από κάποια ουδετερότητα, Οπότε δεν θέλουμε με τίποτα να πάμε να επιβαρύνουμε ακόμα περισσότερο τους ε, φορολογούμενου. γιατί τελικά αυτοί πληρώνουν την νύφη όσον αφορά τι ε, ευρωπαϊκέ πολιτικές και τις ε, εθνικέ πολιτικές. Οπότε βλέπουμε ότι η αρμοδιότητα για τα φορολογικά μένει στα κράτη-μέλη. Οπότε, εάν τα κράτη-μέλη κλείσουν κάποια πολιτική συμφωνία και αποφασίσουν για έναν καινούριο πόρο ή για υπάρχοντες πόρους να τον διαθέσουν κάπου, ε, τότε το περιθώριο λιγμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα είναι όπως έχουν ε, οι τοπικές αρχές για τα φορολογικά. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μεταβίβαση αρμοδιότητας από τα κράτη-μέρη στην κοινότητα. Επεξεργαζόμαστε λοιπόν συνεχώς την, μάλλον, τη μεταρρύθμιση αυτή με βάση ένα σταθερό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι πόροι μας συνάδουν με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Αυτή είναι η βάση η οποία για μας φαίνεται ότι είναι ικανοποιητική δεδομένα των εργασιών μας και το χρονοδιάγραμμα καθώς και οι πολιτικές δυσκολίες που θα έχουμε ενώπιόν μας πρέπει να έχουν μόλις ε, υπενθυμιστεί αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη πράγματι όπως υπενθύμησε ο κύριος ε, Μόντι. Χαιρετίζω τον κύριο Φερχόφστατ Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να φτάσει το εδώ. Κύριε Καλφίν, θέλετε να λάβετε εσείς το λόγο τώρα. Πάρα πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Μόντι, τον πρόεδρο Μόντι, για την πάρα πολύ ικανή προεδρία του της ομάδας μας που έχει τόσο δύσκολο καθήκον. Καταρχήν, τα κάτι μελη συμφώνησαν να συζητήσουν για τον προπολογισμό με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό είναι αυτό, αλλά δεν είναι το άπαν. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και αυτό είναι και το αντικείμενο της πρώτης έκθεσης <clears throat> αξιολόγηση. Υπάρχει ένα συστημικό πρόβλημα του προπολογισμού που δημιουργεί και δημοσιονομικέ εντάσει σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία δημιουργούνται σε ό,τι αφορά την λειτουργία, την ομαλή λειτουργία των ευρωπαϊκών πολιτικών και υπάρχει ένα σύστημα το οποίο το οποίο δεν είναι ούτε δημοκρατικό ούτε διαφανές. Αυτό δείχνει αυτή η πρώτη έκθεση. Τα επόμενα βήματά μας θα πρέπει να κινηθούν προς την κατεύθυνση της θεραπείας αυτών των προβλημάτων. Έχουμε επιχειρήματα πολύ ισχυρά, μερικά από αυτά τα ανέφερε ο κύριος Λαμασούρ. Ο στόχος μας δεν είναι να άρουμε την ε, δημοσιονομική αυτονομία των κρατών μελών. Ούτε θέλουμε να προσθέσουμε πρόσθετο άχθος για τους φορολογούμενους. Αλλά είναι λύσεις που θα κάνουν πιο αυτόνομο τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και θα ε, περιορίσουν τη δυνατότητα λήψης απόφασης των κρατών μελών που κάνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά όμοιρο του εθνικού του προϋπολογισμού με την εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και οι συμβολές στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό είναι πρόσθετο άχθος <clears throat> για τα κράτη-μέλη. Οποιοδήποτε ευρώ δίδεται στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό σε κάποια κράτη-μέλη θεωρείται ότι έχει αφαιρεθεί από τον κοινωνικό τομέα από το επενδύσεων κτλ. Όλα αυτά είναι μια τελείω λανθασμένη αντιμετώπιση βέβαια. Μπορεί να χρειαστούν διαφορετικέ λύσει λοιπόν από ένα κράτο σε κάποιο άλλο, αλλά ο στόχος είναι να παραμείνει η κυριαρχικότητα και η αυτονομία λήψη απόφαση των κρατών μελών. Είναι απαραίτητο να συμμετέχουν όλα τα θεσμικά όργανα σε αυτή τη συζήτηση. Το Συμβούλιο συμφώνησε στο να υπάρξει αυτή η ομάδα εργασίας όχι με μεγάλη ευκολία βέβαια, ήταν τμήμα των τελικών αποφάσεων που ελήφθησαν για το τωρινό πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχει εκπροσώπους στο Συμβουλίο, οι οποίοι είναι εξαίρετοι, αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να έρθει η συζήτηση αυτή με τα επιχειρήματα αυτά στα Εθνικά Κοινοβούλια και στα Εθνικά Όργανα Λήψης Απόφασης που περιλαμβάνει και τις εθνικές κυβερνήσεις. Εμείς μόνο επιχειρήματα μπορούμε να παρουσιάσουμε διαφορετικές προτάσεις, διαφορετικές κατευθύνσεις. Έχουμε συζητήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε συζητήσει και με την Κομισιόν, αλλά τώρα πρέπει να φέρουμε τη συζήτηση στις εθνικές κυβερνήσεις. Αλλιώς τα συστημικά προβλήματα με τον προϋπολογισμό μπορεί να μετατραπούν σε πολιτικό πρόβλημα που θα υποσκάψει και το νόημα της ευρωπαϊκής πολιτικής και των πολιτικών που ασκεί. Πράγματι, λέει ο πρόεδρος Αρτουή, θα πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο τη σχέση μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και έτσι η διακοινοβουλευτική διάσκεψη θα αποκτήσει περισσότερα σάρκα και οστά. Ο κύριος Φερχόφστατ έχει το λόγο. Πάρα πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω και να επιβεβαιώσω αυτά που είπε ο κύριος Λαμασούρ. Ελπίζω ότι ο κύριος Μοντή θα αντιμετωπιστεί με τον ίδιο ενθουσιασμό στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων. Θα τον υποδεχθούν ενθουσιοδός, γιατί εκεί βρίσκεται ο πυρήνας του προβλήματος. Ελπίζω λοιπόν ότι θα γυρίσετε σως και αυλαβείς από τη συνάντηση με την Κορεπέρ είναι πολύ πιο δύσκολη εκεί η συνεργασία από αυτή που έχετε να αντιμετωπίσετε από την Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί η έκθεση αυτή ε, ουσιαστικά απεικονίζει αυτά τα οποία έχει διαπιστώσει και η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο στο παρελθόν σε πολλές ευκαιρίες. Βέβαια η δεύτερη φάση του εγχειρήματο θα είναι πιο δύσκολη γιατί θα πρέπει να γίνουν κάποιες επιλογές. Θα πρέπει να πούμε πρέπει οι πόροι αυτοί να χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφεξής και θα πρέπει να ξεπεράσουμε το τωρινό σύστημα και ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να ξαναγυρίσουμε στην αρχική μορφή χρηματοδότησης της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1957-58. Με την επιστροφή στη Μεγάλη Βρετανία στη δεκαετία του 80 αλλάξαμε το σύστημα και επειδή δεν είχαμε και τα τεχνικά μέσα να έχουμε ένα ενιαίο σύστημα ΦΠΑ, τότε υπήρξαν προβλήματα. Τώρα όμως είναι πολύ πιο εύκολο να εφαρμόσουμε ένα τέτοιο σύστημα σε πραγματικό επίπεδο και όχι μονάχα σε επίπεδο στατιστικών. Θα πρέπει λοιπόν με την επόμενη έκθεση να ξεκινήσει η πραγματική εργασία. Το γνωρίζει και ο πρόεδρος Μόντι ότι τότε λοιπόν θα είναι απαραίτητο να προβούμε σε επιλογές. Το γεγονός όμως ότι υπάρχουν στην ομάδα αυτή οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου και συμμετέχουν και ενέκριναν αυτή την έκθεση, αυτό είναι κάτι το καινοφανές, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί στο παρελθόν, γιατί οι προσπάθειες μας στο παρελθόν, όπως θυμάται ο κύριος ε, Λαμασούρ, δεν ήταν καρποφόρες. Εκφράσαμε απλώς τις απόψεις μας και καταλήξαμε μονάχα σε μια έκθεση των τριών. Είχαμε καταλήξει, έχουμε καταλήξει εδώ τώρα σε μια έκθεση τριών θεσμικών οργάνων και όχι μονάχα κομισιών ή κοινοβουλία. Αυτό ήθελα να υπογραμμίσω. Ευχαριστώ και ο πρόεδρος. Οποιοδήποτε ε, εγχείρημα θα πρέπει να βασιστεί στην σοφροσύνη και στην σοφία της ομάδος αυτής. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους μόνιμους ηγητές, καταρχήν στον κύριο Λεβεντόφσκι. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ καλό το ότι ήρθε με τόσο ενθουσιασμό εδώ ο κύριος Μόντιος πρόεδρος με μια ομάδα που εδώ, αλλά βέβαια είναι και θέμα δικαιοσύνης το, το ότι έχουμε από την άλλη μεριά τον Αλένα Μασούρο στην πολιτική ομάδα, γιατί ανέκαθεν αυτό πρέσβευε τον. Έχουμε μια τέτοια εκβάθρον μεταρρύθμιση των συστήματος των ε, ίδιων πόρων και θυμάται ο Φερχόφστατο τη λογική εκείνη των, των ε, πολυμερών διαπραγματεύσεων και είναι σωστό αυτό να υπάρχει μια τέτοια ζώσα μνήμη των διαπραγματεύσεων και αυτή η έκθεση αποκαλύπτει την αλήθεια, το πώς έχουν τα πράγματα. Κάτι το οποίο βέβαια δεν φέρνει τόση αισιοδοξία ε, όπως είπε στην εισήγηση ο Μάριο Μάντη γιατί απέχουμε πάρα πολύ από την αρχική πρόταση που είχε συζητηθεί τον Ιούνιο του 2011 γιατί είχαμε αυτή την εξέλιξη από πλευρά των δαπανών και ολοκληρώθηκε αυτή η εξέλιξη για τις δαπάνες αλλά πάλι ήταν επαναστατική εξέλιξη όσον αφορά τα έσοδα για, από πλευράς εισόδων για τον ΦΠΑ, από πλευρά συστήματος συναλλαγών, άρα είχαμε για τα λάμψαμς, για τις διορθώσεις. Κάτω από ποσά τέλο πάντων που και αυτό ε, ε, ε τροποποιήθηκε. Οπότε και έτσι ε, είδαμε το πώς έγινε η υλοποίηση αυτής της μεταρρύθμισης γιατί είχαμε πει ότι θα πρέπει η φορολογία να βοηθά τον προϋπολογισμό. Και βέβαια αυτό, σε αυτό ευώθησε πάντα η ενισχυμένη συνεργασία. Άρα, βλέπουμε τώρα τι ευκαιρίες υπάρχουν και τι φραγμοί για να συνεχιστεί αυτή η μεταρρύθμιση και αυτό όμως θα πρέπει να γίνει παράλληλα με το να κτηθεί πάλι η εμπιστοσύνη προς τα ε, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και προς τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. αυτά μεταξύ τους είναι διαχώριστα. Πάνε μαζί, αλλιώς η αποστολή αυτή είναι αδύνατη. Βλέπουμε και τι πρόκειψε από τις ε, ευρωπαϊκέ εκλογέ Δεν ήταν τα πράγματα τόσο, τόσο ρόδινα. Οπότε, καλή τύχη. Νομίζω ότι με αυτή την αναθεώρηση έχει και το Κοινοβούλιο μια ευκαιρία ώστε να διαμορφώσει το γίγνεσαι αυτό. Ο πρόεδρο, ευχαριστώ. Είχαμε ε, πάντω κι άλλον ένα συνεισηγητή εκτό από εσά, τον Ζεραλντεπρέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Μόντι, αναφέρετε πριν λίγο ότι αυτό το έγγραφο είναι το αποτέλεσμα των ε, αποτέλεσμα ε, της ομάδας το οποίο είπατε ότι είναι κάπου ήπιο δεν νομίζω ότι είναι ήπιο ε, ε, αυστηρό, σκληρό είναι και το διάβασα και είδα ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή διανοητική προσπάθεια πάρα πολύ καλά συναρθρωμένο και τεκμηριωμένο πάντως εγώ έχω στρατευτεί υπέρ των ιδίων πόρων όπως πάρα πολύ εδώ στην Επιτροπή μας και δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι αυτός ο λυρισμός με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα πράγματα σήμερα θα είναι πραγματικότητα αύριο. Όταν δηλαδή έχουμε του ίδιους πόρους, κάποια από αυτά που έχουν ζητηθεί στο Συμβούλιο μεταξύ αυτών που θέλουν περισσότερα χρήματα για την Ευρώπη και εκείνων που θέλουν λιγότερα, αν θα είναι δυνατόν αυτή η ζήτηση να γίνει αλλού. Γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι εύκολα δέχονται να ε, γίνει αύξηση ε, στους ίδιους πόρους και άλλοι είναι πιο διστακτικοί. Οπότε νομίζω ότι όταν κάνουμε την αξιολόγηση για τους ε, ίδιους πόρους να ξέρουμε ότι αυτό πρόκειται να έχει επιπτώσεις και εις τον κοινοβουλευτικό διάλογο. Οπότε κάθε φορά που ζητείτε περισσότερο χρήμα από το Συμβούλιο τότε χρειάζεται να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση όσον αφορά το τι ζητάμε από τον πολίτη και τι αποφασίζουμε να έχει ως πόρος ο προπολογισμό. Κύριε Μόντι, θέλω να ρωτήσω το εξή σε σχέση με την ομάδα σας. Εάν κατάλαβα καλά, Πρόεδρε, από το κείμενο σας τώρα πρόκειται να στείλετε κάποια ερωτήματα σε μια ομάδα εμπειρογνωμών. Βλέπω αυτό στη σελίδα 32 και έχουμε μια σειρά ερωτήσεων που θέλετε να τις υποβάλλετε σε εκείνους. Νομίζω ότι ε, κάποια από αυτά τα ερωτήματα δεν είναι θέμα περιγνωμοσύνης, δεν είναι τεχνοκρατικά. Είναι πολιτικά θέματα. Οπότε αυτό και με προβληματίζει. Να, να σας πω κάποια παραδείγματα γιατί νομίζω ότι πρόκειται για ε, πολιτικές επιλογές. Και δεν είμαι σίγουρος ότι είναι δυνατόν αυτοί οι εμπειρογνώμονες έχουν, να βρουν την νομιμοποίηση που χρειάζεται για να απαντήσουν. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο εδώ πέρα το εντοπίζεται εδώ και το οποίο επίση δεν έχει απάντηση εύκολη. Εάν δεν καταλήξουμε πουθενά όσον αφορά του ίδιου πόρου, γιατί το Συμβούλιο δεν έχει δείξει θετική ε, ανταπόκριση σε όλε αυτέ τι απόπειρε, λέτε για την λαϊκή υποστήριξη. Αλλά εν απουσία αυτή τη λαϊκή ε, υποστήριξη για την εξαίρεση του τι θα γίνει, πώς θα, πώς θα αποσπαστεί αυτή η έγκριση η, η λαϊκή. Τι στρατηγική θα μετέλθει κανείς από και τα κράτη-μέλη είναι τόσο δυσταρχικά, ούτως ώστε να έχει κανείς την υποστήριξη του κόσμου για μια τέτοια μεταρρύθμιση όπως θέλουμε να κάνουμε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική ε, αυτή, ε, αυτή η υπόθεση όσον αφορά την αίσια κατάληξη και τη διαδρομή μου. Άλλη μια ερώτηση εγώ για εσά. Από τα συμπεράσματα του εγγράφου. Υπάρχει μια πρωτασούλα εκεί στη σελίδα 36 νομίζω που επίσης με προβλημάτισε. Λέτε. Οι βελτιώσεις του τρέχοντα συστήματος είναι δυνατόν να αναζητηθούν με κάποιο είδους ε, αναθεώρηση της χρηματοδότησης των πολιτικών. Και αν γίνεται, να έχουμε βελτίωση μόνο από την τροποποίηση του συστήματος και μετά λέτε, λέτε, πώς θα μπορέσουμε να μεταρρυθμίσουμε αυτές τις ίδιες πολιτικές που αποφασίστηκαν στα πλαίσια του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Και ρωτάω, Πρόεδρε, Μέχρι πού θα φτάσετε, γιατί με αυτή την ε, λογική δεν είναι θέμα προβληματικής ε, των ίδιων πόρων, αλλά είναι πολύ ευρύτερος αυτός ο συλλογισμός, γιατί πια αμφισβητείτε το modus operandi των ευρωπαϊκών πολιτικών. Θέλετε να φτάσετε μέχρι εκεί ή είναι απλώς εδώ ένα ρητορικό ερώτημα. Σας ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο σε αυτούς ε, <clears throat> μεταξύ ημών οι οποίοι ζήτησαν να εκφράσουν κάποια σχόλια, να θέσουν ερωτήματα στους προσκεκλείς. Ο Σανκά, Μανκά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ανάλυση που μας παρουσιάσατε εδώ. Το έγγραφο αυτό είναι εύστοχο, αναφέρεται στα πραγματικά προβλήματα. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει επαρκείς πόρους για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλες τις στρατηγικές που έχει αναπτύξει. Το είπατε πολύ ορθά ότι οι διαπραγματεύσεις του προϋπολογισμού είναι πολύπλοκες και επεπλεγμένες έγιναν 40 μέρε διαπραγματεύσεων για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Παρά όλα αυτά τα προβλήματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμα αρκετά χρήματα για να τηρήσει τι υποχρεώσει που έχει αναλάβει και που απορρέουν και από τι συνθήκε τη Λισαβόνα. Είχαμε ήδη χθε συναντήσει με τις Εθνικές εθνικά κοινοβούλια, μα λέγανε οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι δήμαρχοι ότι δεν μπορούσαν να πάρουν τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που του είχαν υποσχεθεί και χρειαζόταν να δανειστούν χρήματα από τι τράπεζε δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι τα πράγματα. Πρέπει να φτιάξουμε ένα πιο ευφυή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα δίνει περισσότερα χρήματα για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τις επιδιώξεις μας χωρίς να επιβαρύνουμε τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περαιτέρω. Αυτή τη στιγμή οι πολίτες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες επομίζονται όλο το βάρος του προϋπολογισμού οι πολίτες μας δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί γίνεται κάτι τέτοιο. Αρχίζουν να, να έχουν την εντύπωση ότι εμείς όλο και περισσότερο παίρνουμε χρήματα από την δική τους τσέπη, από τους εθνικούς προϋπολογισμούς και γι' αυτό υπάρχει φόβος να μην υποστηρίξουν την πρότασή μας. Χρειάζεται μια κοινή αντιμετώπιση και χρειάζονται περισσότεροι πόροι στον κοινό μας προϋπολογισμό. Και σήμερα θα πρέπει να ψηφίσουμε για την αιτήσια επισκόπηση ανάπτυξης για το 2015 υπάρχουν κάποιες, κάποια σενάρια, κάποιες ιδέες που υπάρχουν ήδη στο έγγραφο αυτό. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τη συζήτηση για τους ίδιους πόρους. Εγώ χαιρετίζω αυτή τη συζήτηση για τους ίδιους πόρους, αλλά νομίζω πρέπει να περιοριστούμε σε ορισμένες αρχές. Μία από αυτές πρέπει να είναι ότι η μεταρρύθμιση αυτή δεν πρέπει να αυξήσει το συνολικό φορολογικό βάρος. Δεύτερη αρχή είναι ότι οι συνεισφορές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό δεν θα πρέπει να κάνουν διακρίσεις εναντίον συγκεκριμένων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τις δραστηριότητες των εταιριών που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί που την χάνουν περισσότερων διακρίσεων στον τομέα του ΦΠΑ δεν θα πρέπει να επηρεαστούμε από μια τέτοια μεταρρύθμιση όπως γίνεται τώρα. Και επίση οι δαπάνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνδέονται με τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να πηγαίνουν στου τομεί αυτού, όπου μπορεί να προκύψει σαφής προστιθέμενη αξία και είναι πιο ουσιαστική η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από ότι η εθνική. Ξέρω ότι υπάρχουν εμπειρογνώμονες, εμπλέκεται και η Ευρωπαϊκή ε, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και οι εμπειρογνώμονες έχουν δηλώσει την πεποίθησή τους ότι υπάρχουν πολλές φορές ε, διακρίσεις αντικές εναντίον εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον εταιριών σε τρίτες χώρες γιατί οι αλυσίδες τροφοδοσίες των επιχειρήσεων αυτών <clears throat> υπάρχουν τα προβλήματα της, ε, του συστήματος για την ε, εμπορία εκπομπών και του, τα προβλήματα ενέργειας τα οποία βαρύνουν περισσότερο τις εταιρείε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε μια ισοδίκια μορφή ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω και οι εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να άρουμε τις διακρίσεις εναντίον των βιομηχανιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην παγκόσμια αγορά. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής, κύριε Πρόεδρε, <clears throat> ο κύριος Δελάνο. Αν δεν βρούμε λύση για αυτά τα προβλήματα των ιδίων πόρων, εγώ θα ευχηθώ καλό κουράγιο σε αυτούς οι οποίοι θα εκτεθούν στην επόμενη προεκλογική εκστατεία για τις ευρωεκλογές. Γιατί οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν μια πιο ορατή, μια πιο αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτά απαιτούν κονδύλια, χρήματα. Λάθος είναι να μπαίνουμε σε ένα σύστημα το οποίο δεν τα αποδίδει αυτά. Προφανώς χρειάζονται, χρειάζεται ομοφωνία των κρατών μελών για να τροποποιηθεί το σύστημα χρηματοδότησης. Αλλά θα ήταν χρήσιμο για τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν τους πόρους που χρειάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί εδώ πέρα είμαστε κολοβωμένοι κατά κάποιο τρόπο. Μπορούμε να ψηφίσουμε τις δαπάνες αλλά όχι τα έσοδα. Το να θεωρούμαστε λοιπόν συνομοθέτες στον τομέα του προϋπολογισμού δεν ευσταθεί. Γιατί ελέγχουμε μονάχα το ένα σκέλος του προϋπολογισμού που είναι οι δαπάνες. Χρειάζεται σήμερα μια πραγματική πολιτική θέληση για να αλλάξει αυτό. Πρέπει κάποια στιγμή όμως να τονίσουμε την πολιτική μας θέληση να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Είναι πολύπλοκες βέβαια οι λύσεις και δεν θα μπορούσαν να συμφωνήσουν όλοι πώς θα γίνει κάτι τέτοιο. Μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε το, ένα σύστημα συνολικό ΦΠΑ το οποίο θα είναι ε, για όλους. Αλλά υπάρχουν άλλοι φόροι που ζητούν ορισμένοι φόροι ενέργειας, φόροι χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που θίγουν περισσότερο ορισμένε χώρες. Εδώ θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα και να δούμε πώς θα είμαστε πραγματιστικές για το σύστημα ε, ιδιών πόρων, το σύστημα του παζαριού που έκανε η κυρία Θάτσερ δεν μπορεί να συνεχιστεί πλέον. Είναι απόλυτα απαράδεκτη η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και πρέπει να βρούμε λοιπόν ένα άλλο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε τη χρηματοδότηση του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος Τάγκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ κύριε Μόντε και τα μέλη της ε, ομάδας που βρίσκονται εδώ της ομάδας υψηλού επίπεδου. Φυσικά η Επιτροπή μας ε, ανυπομονεί, αδειμονεί. Αλλά εντάξει, όπως είπατε, είναι άχρωμη η έκθεση αυτή, τι να κάνουμε. Um, Δέχομαι ωστόσο ότι επιλέξετε την προσέγγιση αυτή όπως εξηγήσατε. Αυτή την ευρεία προσέγγιση χρειάζεται μια ευρεία προσέγγιση, μια κοινή ανάλυση του προβλήματος. Ιδάλως ανακύπτεται το θέμα δικαιοσύνης και ισότητας. γιατί οι ίδιοι πόροι πάντα θα οδηγούν σε φορολογική βάση και αυτό πάντα θα θέτει θέμα δικαιοσύνη και ισότητας. Και φυσικά τύφεται και το θέμα των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και μένα με εξέπληξε, με σόκαρε η έλλειψη γνώσεων για το θέμα από το κοινοβούλιο μου, από τον υπουργό μου τον ίδιο. Αυτή η ευρεία προσέγγιση όμως το έθεσε και ο συνάδελφο το ερώτημα αυτό. Έχω δύο ερωτήσει να σα κάνω με τα συμπεράσματα. Εκεί που αναφέρεται ότι υπάρχει σύνδεσμος, σχέση, μια ρητορική ερώτηση κατά πόσο πρέπει να μιλήσουμε για τα έσοδα ή για τις δαπάνες. Ρητορικό το ερώτημα μου φαίνεται. Αυτό τι σημαίνει ότι δεν θέλετε μόνο να εξετάσετε τη χρηματοδότηση των πολιτικών αλλά και τις πολιτικές της ίδια. καταλαβαίνετε ότι θέλετε μια ευρεία προσέγγιση αλλά μήπω ανοίγουμε και το κουτί τη Πανδώρας. Κάτι άλλο που είναι κρίσιμο. Οποιοδήποτε χρηματοδοτικό σύστημα πρέπει να είναι συνεπές. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχει το προπολογισμό μας τώρα. Είναι υπερβολικά εύκολο για τα κράτη-μέλη να λένε ναι, αλλά να πράττουν όχι. Αυτό έχει να κάνει με το ξεχωριστό σύστημα πληρωμών και δεσμεύσεων. Δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα χρονικής συγκυρίας και νομίζω ότι είναι κρίσιμο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόμασταν σε αδίέξοδο με τις πληρωμές. Ακόμα και η Επιτροπή έλεγε ότι πρόκειται για κρίση αλλά θεωρώ ότι είναι κρίσιμη σημασία να υπάρχει ένα χρονικά ορθό σύστημα προπολογισμού προκειμένου να λειτουργεί το ίδιο το σύστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζάνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε για τον ε, πρόεδρο Μόντι αλλά για την ε, ομάδα του για το έργο του. Όπως είπαμε πρόκειται για μεγάλου ελληνικού ε, έργο. Δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο θέμα. Είναι χρήσιμο απολύτως και ελπίζουμε ότι τα επόμενα βήματα πρόκειται να γίνουν ε, με ρυθμό ταχύ και να μας οδηγήσουν σε κάποιες τέτοιες προτάσεις γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Θέλω τώρα να ξεκινήσω με κάτι το οποίο συμφωνώ ε, και το είπε ο κύριος Λαμασούρ και αφορά τους ιδίους πόρους του προϋπολογισμού. Εδώ διακυβεύονται τα πάντα. Η ίδια η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν αποτύχουμε, τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δώσουμε εξηγήσει στον κόσμο. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε πόρους για να χρηματοδοτήσουμε τον προϋπολογισμό. Και τα σημερινά πολύ σοβαρά προβλήματα, τα προβλήματα των πληρωμών, πρόκειται να παροξυνθούν και θα μας οδηγήσουν σε κατάρρευση. Ελπίζω ότι τα κρατη θα καταφέρουν να συμφωνήσουν όσον αφορά αυτήν όλη τη θεματική και το λέω έτσι γιατί ακόμα δεν έχουν συμφωνήσει τίποτα γιατί βλέπω εδώ στο ιστορικό του Κοινοβουλίου ευρεία πλειοψηφία σε σχέση με το ότι θα πρέπει να αποκτήσει ο προϋπολογισμός τους ίδιους πόρους ε, είτε μέσω του, του, φόρου του διοξιδίου, με, με κάποιο φόρο τέλο πάντων. Όμως, όμως, τα κράτη-μέλη ακόμα διστροπούν και αυτό το είδαμε στα πλαίσια του φετινού προϋπολογισμού όπου είχαμε πόρους για το 2014 αλλά τα κράτη-μέλη αποφάσισαν να πάρουν πίσω τα χρήματά τους και να μην λύσουν το πρόβλημα. Και γι' αυτό και είχαμε το πρόβλημα των πιστώσεων πληρωμών. Επίσης πάρα πολύ συμφωνώ ότι όχι μόνο τα κράτη-μέλη, αλλά και εμείς θα πρέπει να δώσουμε το θετικό μήνυμα και να κάτσουμε και να προβληματιστούμε σε σχέση με το τι θέλουμε να γίνει για έσοδα και δαπάνες. Να δούμε και να δουλέψουμε σκληρά, να, κάνουμε, να κάνουμε μια ανάλυση αυτών των δαπανών που, για τα οποία δεν, δεν απαιτούν, δεν, δεν επαρκούν τα έσοδα. Ε, έχουμε πρόβλημα και αυτό το ξέρουν πολύ καλά από την Ιταλία, αλλά δεν είναι μόνο η Ιταλία αυτό ο οποίο δεν χρησιμοποιεί αποτελεσματικά του πόρου. Οπότε, πριν κάτσουμε και ψάξουμε ιδίου πόρου για έσοδα, α κάτσουμε να σκεφτούμε τι γίνεται με τι δαπάνε. Να δούμε πώ θα ε, πώς, πώς τα χρήματα εάν φτιάχνουμε μια προσθεμένη αξία ε, στα κράτη-μέλη και έτσι θα πρέπει να έχει μια προσθεμένη αξία που φτιάχνει ο ευρωπαϊκός προπολογισμό. Αλλιώς κανένα κρατός μέλος δεν θα θέλει να δώσει ε, πόρους στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Και, εν κατακλείδη, ένα τελευταίο θέμα όσον αφορά τις ε, προτάσεις για τον ε, φόρο των συναλλαγών, για τον φόρο του διοξιδίου, υπέροχες ε, προτάσεις. Ναι, έξυπνη πρόταση, αποτελεσματική αυτή η φόρη και αν το χρησιμοποιήσουμε πρόκειται να αναβληθεί η μετακύληση του βάρους και του άχθους στους πολίτες. Γιατί είδαμε τι γίνεται με την χρησιμοποίηση του ΦΠΑ. Γιατί ακόμα και κατά μία μονάδη αύξηση του ΦΠΑ είναι κάτι πολύ βαρύ. Και είδαμε, μπορούμε να οδηγηθούμε επίσης την άλλη μεριά σε ε, βλάβη του περιβάλλοντος σε σχέση με το πώς χρησιμοποιείται ο φόρος του διοξιδίου. Άλλη τώρα πρόταση θα μπορούσε να είναι να μελετηθεί το πώς να εισπράξουμε κάποιους πόρους για τον προϋπολογισμό φορολογώντας κάποιες δραστηριότητες οι οποίες σήμερα είναι παράνομες. Κάποια έχουν νομιμοποιήσει κάποιες δραστηριότητες όπως ελαφρά ναρκωτικά, πορνεία, οπότε να το παράδειγμα το πράγμα το παίρνω από κάποιες πολιτείες αμερικανικές, οι οποίες πολιτείες έχουν νομιμοποιώσει τα ελαφρά ναρκωτικά. Το κάνουν κάποια κράτη-μέλη. Το χρησιμοποιούν σε επιχείρημα. Επίσης είναι σημαντικό να δούμε πώς θα έχουμε την τροφοδότηση από τους ιδίους πόρους και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε το συντομότερο δυνατόν. γιατί η ρεφιοκρατία στην Ευρώπη λειτουργεί με βραδίτητα. Όμως θα διακυβεύουμε την αξιοπιστία μας. Διακυβεύουμε τις επενδύσεις. Αλλά να, η πρώτη και καλύτερη επένδυση είναι ο προπολογισμό. Επομένω, να, γιατί πρέπει να δουλέψουμε προ αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εσά Πρόεδρε Μόντι για την ομάδα εργασία για το έργο που σήμερα μας παρουσιάσατε. Ε, συμφωνώ με αυτό που είναι που έλαβε το λόγο προηγουμένως. Αυτό το ζήτημα δεν ε, είναι πολύ συγκεκριμένο γιατί μπορεί να φτάσει ε, και να επηρεάσει όλο το ευρωπαϊκό τοπίο. Επομένως είναι πολύ σημαντικό χρειάζεται μια αποφασιστική πολιτική. Γιατί με αυτή την ομάδα υψηλού επίπεδου πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία όπως θυμάστε είχε γίνει αυτό σε Συμβούλιο και Επιτροπή κατά την προηγούμενη θητεία για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και έχει επιπτώσεις στην ζωή των Ευρωπαίων γιατί αφορά την φορολόγηση. Είναι πολύ βασικά ε, θέματα αυτά στην ε, συγκρότηση ενός κράτους στο δυτικό κόσμο. Οπότε το έργο το οποίο πρέπει να επιτελέσουμε και εμείς και εσείς χρειάζεται θάρρος, χρειάζεται φαντασία. Ακούσαμε τι είπε και ο τελευταίος προλαλής σας. Οπότε φαντασία και θάρρος χρειάζεται. Οπότε, όπως είπατε πρόεδρε, ακόμα το τοπίο είναι ασαφές, γκρίζο σήμερα. Άρα χρειάζεται να προσπαθήσει κανείς ε, με ακρίβεια, ενδελεχώς και θα πρέπει να κάνει έργο μακρόπνοη. Οπότε και στο Κοινοβούλιο και στην Ευρώπη. Βρισκόμαστε σε σημαντική συγκυρία, έχουμε την ευελιξία, έχουμε το ε, πρόγραμμα Juncker και όλα αυτά κάποιοι λένε ότι δεν επαρκούν. Πάντοτε αναζητούμε το καλύτερο. Δεν μου αρέσουν αυτές οι προοπτικές, αλλά θα πρέπει να βρούμε τελικά τη λύση και να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη της Ευρώπης. Και αυτό να γίνει εκτός και άσχετα με τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Έχω σύντομες ερωτήσεις, τρεις. Για να καταλάβουμε πώς θα πρέπει να εργαστούμε για να προχωρήσει η υπόθεση. Πρώτα-πρώτα. έτσι τις εκτιμήσεις Θεωρείται ότι πέραν αυτών που, των δεδομένων που έχει ότι θα μπορέσουν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να καταλήξουν σε ένα καινούριο σύστημα ιδιών πόρων μέσα στα όρια και στα πλαίσια της ε, εντολής αυτής της θητείας. Τι λέτε, δεύτερη ερώτηση. Ποια κράτη-μέλη δείχνουν περισσότερο πνεύμα συνεργασία σήμερα και θα μπορούσαν να είναι σε εισαγωγικά οι σύμμαχοι σε αυτό το έργο που έχουμε αναλάβει. Τέλος, από πλευράς μεθοδολογίας της ομάδας υψηλού επίπεδου που διευθύνεται. Όπως είπατε, πότε θα αρχίσει το γκρίζο έγγραφο να αποκτά χρώματα. Πότε θα καταλήξετε σε κάποιες προτάσεις που εμείς θα μπορέσουμε να τις υλοποιήσουμε, να τις συζητήσουμε, προτάσεις με τις οποίες θα μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο. Πώς φαντάζεστε να καταλήξει αυτό το έγγραφο πέραν του στενού περιεχομένου, αυτό το οποίο θα παρουσιάσετε το 2017. Μονάχα μία διευκρίνηση. Πρέπει ο πρόεδρος Μόντι να φύγει στις 11. 11 και 5 το πολύ, αλλά όχι παραπάνω. Αν θέλετε να απαντήσει όλα τα ερωτήματα αυτά, παρακαλώ να είστε πάρα πολύ συνοπτικοί και σύντομοι. Ο κύριος Μαραγάλο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μόντι για την έκθεσή του. Όπως ελέγχθη πράγματι, φαίνεται ότι αυτή η έκθεση είναι ένα σημείο εκκίνησης, φαίνεται ότι είναι απόλυτα ενημερωμένη και πλήρης και η έκθεση αυτή φυσικά πρέπει να τύχει περαιτέρω εξέλιξης και αντιμετώπισης και υπάρχει τώρα και το στοιχείο του κινδύνου. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να επιλέξουμε και αυτό μπορεί να έχει κάποιο κίνδυνο. Θα πρέπει να καθορίσουμε σαφείς στρατηγικέ με την πεποίθηση ότι πρέπει να βρούμε μια ευρωπαϊκή λύση. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα παιχνίδι όπου εμπλέκονται τα κράτη-μέλη και ο καθένας προσπαθεί να πετύχει να πάρει τα περισσότερα δίνοντας τα λιγότερα. Δεν είναι καινούριο αυτό το παιχνίδι. <clears throat> Πάντα είναι οι πιο ισχυροί εναντίον των πιο αδυνάτων. Οι ισχυρές χώρες είναι αυτές οι οποίες καθορίζουν τη δομή και την ε, λειτουργία του προϋπολογισμού και το θεωρούν σχεδόν φυσιολογικό να εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις αυτές. Αυτό το οποίο δεν πρέπει να δεχτούμε είναι το παιχνίδι αυτό να φέρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα επίπεδο καθημερινής επιβίωσης μονάχα και ανικανότητος να πληρώσει τους επιστήμονες, τους φοιτητές, τις επιχειρήσεις που εκτελούν σχέδια για λογαριασμό τους. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα συλλογικό κινησμό για τον οποίο είμαστε όλοι υπεύθυνοι, ακόμα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρά το γεγονό ότι εμεί είμαστε οι πιο ενεργοί στο να καταγγέλουμε αυτή την ε, κατάσταση. Αλλά ίσω δεν κάνουμε τι απαραίτητε ενέργειε για να αποτρέψουμε. Μέσα στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, ο κινησμό έχει συμπεριλάβει και την έννοια των ιδίων πόρων. Πρέπει να λέμε πόροι των κρατών μελών, γιατί δεν έχουν πια ευρωπαϊκό χαρακτήρα, έχουν μόνο εθνικό χαρακτήρα. Τα πάντα είναι εκτός από ευρωπαϊκή αυτή η πόρη. Ο καλύτερος τρόπος να σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο λοιπόν είναι με το να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πραγματικά ευρωπαϊκούς και ίδιους πόρους. Αυτό σημαίνει μεταρρύθμιση του συστήματος. Χρειάζεται να εισαγάγουμε νέες ιδέες, νέες μορφές φορολογίες οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους την ανάγκη να υπάρξει πόρος ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη απλώς να συλλέγουν, να καταγράφουν αυτή τη φορολογία, αλλά όχι να είναι αυτοί οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες αυτών των πόρων. Κλείνοντας λοιπόν κύριε Μόντι, θέλω να πω ότι ελπίζω θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε θετικά προς την κατεύθυνση αυτή με την Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου και η εντολή της ομάδος υψηλού επίπεδου είχε την ιδέα <clears throat> της λογοδοσίας, της δικαιοσύνης και της διαφάνειας και επίσης εγώ τονίζω την ανάγκη να έχει δημοκρατική νομιμοποίηση. Το νέο σύστημα θα πρέπει να έχει νομιμοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μπορούμε να μείνουμε όμοιροι του ευρωσκεπτικισμού. Δεν μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις για το μελ γνώμονα το πώς θα λειτουργήσει ο ευρωπαϊκός πατριωτισμός σε εθνικό επίπεδο ή αν θα τροφοδοτεί το σκεπτικισμό. Πρέπει να είμαστε γενναίοι, πρέπει να είμαστε πραγματικοί Ευρωπαίοι και πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να έχουμε το θάρρος για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε ένα σύστημα πραγματικό που θα δίνει πόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Κυρία Γη, Γέντα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την παρουσίαση και σας, σας εγχαίρω για το έργο σας. Έχετε εργαστεί πολύ σκληρά Νομίζω ότι ο προηγούμενη ομιλητής έθεσε κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι τι είναι ουσιαστικά οι ίδιοι πόροι. Γιατί ενδεχομένως υπάρχει κάποια σύγχυση στα καρδιμέλια, τι είναι. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποιο δημόσιο φόρουμ να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί προφανώς θα επηρεάσει το φορολογούμενο στην κάθε χώρα και είναι κρίσιμο να κοιτάξουμε το θέμα των εσόδων, ε, του ε, συσσωρευμένου χρέους και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά θα έπρεπε ίσως να συζητηθούν όλα αυτά στο ευρύτερο πλαίσιο του που, προς τα που κινούμαστε οικονομικά. Κοιτώντα το σχέδιο Γιούγκερ και το καθεξής, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει εναρμονισμένη γραμμή σκέψη για το πώς θα επιδράσει και η πολιτική για τους ίδιους πόρους. Είναι τόσο θέμα ταμπού το θέμα των ίδιων πόρων για πολλά κράτη-μέλη. Οπότε θα πρέπει πραγματικά να βρούμε λύσεις που δεν υπάρχουν. Όταν τις βρείτε λοιπόν να μας ενημερώσετε. Ευχαριστώ. Λαμβάνω και εγώ το λόγο τελευταίο ε, ομιλητής. Φυσικά οι ήδη πόροι πρέπει να μας επιτρέψουν να πληρώσουμε τα οφειλόμενα που συσσωρεύονται αυτή τη στιγμή, αλλά οι ίδιοι πόροι θα πρέπει επίσης και για τον απλό φορολογούμενο να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρξει αύξηση του βάρους. Οποιοςδήποτε ευρωπαϊκός ε, <clears throat> φόρος θα πρέπει να σημαίνει μείωση των εθνικών συνεισφορών. Δεύτερον, βρισκόμαστε σε μια φάση παγκοσμιοποίησης. Οποιαδήποτε φορολογία που βαραίνει την παραγωγή θα οδηγήσει σε μετακίνηση επιχειρήσεων και απασχόληση. Αυτά είναι τα μόνα σχόλια που θέλω να κάνω. Έχετε για τα 8 λεπτά που μας μένουν το λόγο κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη της Επιτροπής που πήραν το λόγο και μας έκαναν ερωτήσεις και σχόλια να εξηγήσω κάποια γενικά ζητήματα τα οποία ακούσαμε εν συντομία, αλλά φυσικά κάθε παρέμβαση τα ληφθεί υπόψη σοβαρά, θα εξεταστεί υπό επισταμένος και θα τα λάβουμε υπόψη αυτά για τις περαιτέρω σκέψεις μας. Αρκετοί από εσά ε, υπογραμμίσατε την ε, θεμελιώδη φύση του ζητήματο αυτού. Είπατε ότι αυτό αποτελεί πράξη ιδρυτική για το Κοινοβούλιο. Όντως, εδώ αγγίζουμε ένα θέμα το οποίο έχει μία σημασία που συνδέεται με την ταυτότητα, την ιστορία, την ίδια τη θεσμική φύση και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα εκ παραλλήλου να διασκεδάσω τον ενθουσιασμό από δικής μας οπτικής πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουμε να τα θέσουμε αυτά ως ένα καθαρό όφελος στο το σύστημα για λόγους διπλωματίας και θεσμικής ισορροπίας. Καταλαβαίνω όμως ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να είναι οι πιο άμεσα εμπλεκόμενοι για την ανάπτυξη των νέων αυτών προοπτικών. Οι τρεις μου συνάδελφοι από την ομάδα, ο κ. Λαμασούρο, ο κ. Καλφίν και ο κ. Βερχόφστατ, ανέφεραν στοιχεία με τα οποία ασφαλώς ε, συμφωνώ απόλυτα. Κάποιοι από αυτούς είπαν και συμφώνησαν και άλλα μέλη της Επιτροπής ότι σε τελική ανάλυση θα πρέπει σε κάποιο βαθμό να επανέλθουμε σε ένα σύστημα το οποίο ήδη υπήρχε στα δεκαετία του 50, του 60 Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, αν και όχι φωναχτά, όλοι σε επίπεδο ευρωπαϊκό και εθνικό, εθνικών κρατών μελών, βρισκόμαστε σε φάση διαφορετικών μεταρρυθμίσεων. Αυτό σε κάποιο βαθμό αποτελεί μια άσκηση αντίθετη προς τις μεταρρυθμίσεις. Γιατί το περσινό έτος περιλαμβάνει κάποια στοιχεία τα οποία ήταν πιο καλά δομημένα και που έφτιαχναν ένα σύστημα καλύτερο από αυτό που ακολούθησε. Αυτό, αυτή η εικόνα της κυρία Θάτσερ ασφαλώς πληρεί τις προϋποθέσεις της ισότητας των φύλων. Δεν θα θέλαμε όμως να αυξηθεί το επίπεδο δυσκολίας σε επίπεδο 28. Um, Να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τους δύο μόνιμους εισηγητές, τον κύριο Λεβαντόφσκι, τον οποίο ευχαριστώ και ιδιαιτέρως για την αρχική συμμετοχή στην ομάδα ως εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου της Επιτροπής, συγγνώμη. Και τον κύριο Ντεπρέ, ο οποίος έθεσε τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Αν σωστά κατάλαβα, δεν κατανοεί κάποια από τα ερωτήματα που θέτουμε στους εμπειρογνώμονες, γιατί θεωρεί ότι είναι ερωτήματα πολιτικής φύσεως. Κύριε Ντεπρέ, έχετε αντιληφθεί ακριβώς ποια είναι η χρήση και η αξιοποίηση των εμπειρογνωμόνων. Πιστεύαμε ότι δεν υπήρχε πραγματικά λόγος να αναζητήσουμε εμπειρογνωμοσύνη επί των συγκεκριμένων τεχνικών λύσεων που θα μπορούσαν να δοθούν σε θέματα ίδιων πόρων τα συν, μείον κτλ. Έχουμε δικός μας ε, εμπειρογνώμονες, τεράστια εμπειρογνωμοσύνη σε όλα τα θεσμικά όργανα. Άρα, το πρόβλημα, αν εξετάσουμε τι έχει γίνει στο παρελθόν, τα προβλήματα και τα αδιέξοδα δεν προέρχονταν από την φορολογική εμπειρογνωμοσύνη. Αλλά προφανώς, αν οι περασμένες προσπάθειες ε, συστηματικά αποτύχαναν, αυτό πρέπει να οφειλόταν σε άλλους λόγους. Και γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ με όλους εκείνους που μίλησαν ε, για ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο χρειάζεται στην αξιολόγησή μας και στην εξέτασή μας. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να καταλάβουμε σε λεπτομερές επίπεδο τι προκάλεσε το αδιέξοδο στην πολιτική μέθοδο, στην ε, στρατηγική μέθοδο κατά το παρελθόν. Γι' αυτό λοιπόν όταν ε, κάναμε διαγωνισμό για τους εμπειριαγνώμονες στους ε, όρους του διαγωνισμού συμπεριλάβαμε και τα πολιτικά αυτά τα στοιχεία, τις πολιτικές αυτές γνώσεις. Αυτό μου θυμίζει κάπως το έργο που έκανα για τον πρόεδρο Μπαρόσο το 2010 για την ενιαία αγορά. Υπάρχουν αμέτρητες εκθέσεις που παρουσιάζουν το τι γίνεται για να ολοκληρωθεί η νέα αγορά, για να είναι πιο ζωντανή κτλ. κτλ. Δεν είναι όμως ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι να κατανοήσουμε το γιατί, γιατί δεν εφαρμόστηκαν κάποιες προτάσεις, γιατί δεν αποφασίστηκαν. Και εδώ λοιπόν κάτι παρόμοιο συμβαίνει. Και γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζουμε το γεγονός ότι τα θεσμικά όργανα μας έδωσαν ε, τη σύνθεση των ομάδων που είναι πολύ πολιτική ασφαλώς, ιδιαίτερα πολιτικός, πολιτικό πνεύμα. Και γι' αυτό λοιπόν αναζητούμε τεχνογνωσία. Όσο για το ευρύτερο πλαίσιο. Δεν θέλουμε να ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας, όπως είπε ο κ. Και όταν επιλέγει κανείς μια ευρύτερη προσέγγιση, πάντα έχει το πρόβλημα κανείς των ορίων. Ιδάλλως γίνεται καταντάει κανείς στην κυκλοπαίδεια και είμαστε σίγουροι ότι κανείς δεν πρέπει να ακολουθήσει τις συστάσεις του. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να μας λάβουν στα σοβαρά και τις προτάσεις μας αν ακολουθήσουμε δύο λέξεις κλειδιά. Πολιτικοποίηση Go back again to one concrete experience many, many years ago. Και εξέταση όλων αυτών σε ένα πακέτο ενδεχομένω, σε μία δέσμη. Να σας μιλήσω λοιπόν και πάλι όταν ήμουν το 96-97 και ξεκίνησα το έργο μου στην Επιτροπή για τον Φορολογικό Συντονισμό. Και αυτό ήταν αδύναμο, αδύνατο έργο. Γιατί κατά τα άλλα δεν είχε κανένα ενδιαφέρον, για να σας πω με πάσα ειλικρίνεια. Ο τρόπος με τον οποίο μετατρέψαμε λοιπόν το αδύνατο σε συγκεκριμένο ψήφισμα του Συμβουλίου 1η Δεκεμβρίου 1999 για να την αντολογία για την εταιρική φορολόγηση και με την ε, βασικές αρχές για τις ε, αποταμιεύσεις ήταν με το να κάνουμε το θέμα αυτό να δώσουμε την πολιτική χρειά στο θέμα αυτό. Πιέσαμε τους ε, Υπουργούς Οικονομίας και τελικά ήρθαν σε δύσκολη θέση. Ήσασταν ε, κι εσείς ε, Υπουργός Οικονομίας τότε. Γιατί οι Υπουργοί, όπως και οι αρχηγοί κυβερνήσεων, μιλούσαν καθημερινά για την ανάγκη υποστήριξης της απασχόλησης και λέγαμε «Ναι, αλλά όσο αφήνουμε αναξέλεκτο το φορολογικό σύστημα και έτσι το φορολογικό βάρος του κεφάλαιο και στις ε, ε, εταιρείε μειώνεται και η συνεργασία αυξάνεται διαρκώς, ουσιαστικά κάνετε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που διακηρύσσετε καθημερινά. Αποφάσισαν λοιπόν να το αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό. Η άλλη καλή ιδέα ήταν να μπει ένα πακέτο προκειμένου να έχει κάθε χώρα και την πικρή αλλά και τη γλυκιά διάσταση του μέτρου. Δεν θέλω να τα υπεραπλουστεύσω αυτά. Αλλά νομίζω ότι κάθε εμπειρία, ακόμα και παραμικρή, μας προσφέρει ένα μήνυμα, ένα, μια εμπειρία. Ύστερα, η υποστήριξη από πλευρά του κοινού, πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση ασφαλώς. Πιστεύω όμως ότι ένα τμήμα του εγχειρήματο. όχι τόσο θετικό για τους φορείς της ε, Ευρωπαϊκής Διαδικασίας θα είναι το να αποκαλύψουμε κάποιες ασυνέπειες. Κάποιες ασυνέπειες ε, σε ό,τι αφορά και τα χρονικά το χρονικό χρονοδιάγραμμα, όπως είπε ο κύριος Τάγκ. Όπως είπατε και εσείς κύριε Τάγκ, ότι άλλο λέμε και άλλο κάνουμε. Λέμε ναι και λέμε και κάνουμε όχι. Δεν θα δραπούμε να επισημάνουμε με κάθε σεβασμό περιπτώσεις όπου αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Και εν συντομία. για την ε, αίτηση να υπάρξει ένα ευρύτερο πλαίσιο. Όλοι σας νομίζω έχετε υποστηρίξει αυτή την άποψη και η η κυρία Ριάντα τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ευρύ πλαίσιο στην οικονομική με την οικονομική έννοια στην τωρινή οικονομική κατάσταση και πόσο ο προϋπολογισμός και οι ήδη πόροι θα πρέπει να συνδεθούν με το γενικό οικονομικό πλαίσιο και την συγκυρία τι ρόλο θα μπορούσαν να έχουν σε αυτή την ε, κατάσταση της κρίσης. Κύριε Μαραγκάλ, το να έχετε νομιμοποίηση αυτό θα είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό όμως πιστεύω ότι σε τελική ανάλυση η έκθεσή μας θα πρέπει να απευθυνθεί όχι μόνο στα ευρωπαϊκά όργανα, αλλά σε μια πιο αναγνώσιμη μορφή, αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, προς τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ώστε να καταλάβουν τι εμπλέκεται εδώ και τι διακυβεύεται. Και για να αποφύγουμε ότι τα μόνα πράγματα που θα ακούν είναι αυτά που τους λένε οι εθνικές αρχές που τις σέβομαι πάρα πολύ όπως ξέρετε πάντα ο κύριος Ζάνη και ο κύριος Βιώτη. Με διαφορετικό τρόπο και οι δύο είπαν ότι πρέπει να είμαστε εφάνταστοι στο έργο μας αλλά και τολμηροί και ελπίζω ότι δεν θα μας λείψει τη μία ούτε θα πρέπει να κάνουμε κάποια ανάλυση των ε, δαπανών κύριε Ζάνη. Δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο και να δώσουμε την ε, εντύπωση ότι θέλουμε να παραταθεί η εντολή μας ούτως ώστε να πούμε τη γνώμη μας για, για θέματα για τα οποία κανένας δεν μας ρωτάει. Ταυτόχρονα όμως κάνουμε το καθήκον μας όσον αφορά το να φτάσει η ανάλυση μας εκεί που χρειάζεται ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες λογικές και εις βάθος και πιστικές απαντήσεις όσον αφορά το πρόβλημα της, ε, των ιδίων πόρων. Όχι, δεν θέλουμε να γενικολογήσουμε πάρα πολύ, αλλά το θέλουμε και να είμαστε πάρα πολύ στενά τεχνοκρατικοί για τους ίδιους πόρους. Κύριε Βιώτη. Όντως, κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα, οπότε και θα ε, δώσουμε χρώμα σε αυτό το έγγραφο που τώρα είναι ή μαύρο και οι προτάσεις μας θα συνταράξουν. Γιατί τελικά η εύκολη συμφωνία όταν κανένα δεν θέλει να παραχωρήσει τίποτα που να παραβλέπει τον εαυτό του και να ωφελεί όλου του άλλου. Εγώ πάντω θα προβληματιστώ πάρα πολύ για τη δεύτερη ερώτησή σα όσον αφορά το ποια είναι τα κράτη τα οποία μπορώ να φανταστώ ότι θα συνεργαστούν πιο πρόθυμα μαζί μα. Οπότε δεν μπορώ τώρα ευθύ αμέσω να σα ε, απαντήσω. Μια ώρα πριν πάω στην Κορεπέρ. Δεν θα ξεχάσω όμω αυτό που ρωτήσατε στα Κύριε Πρόεδρε, έλαβα πολύ σοβαρά υπόψη αυτό το οποίο είπατε και επίσης ε, συμφωνώ με την ε, οπτική γωνία. Την οικονομολογική με την οποία ξέρετε ότι ε, δρώ και εγώ τα τελευταία χρόνια και συμφωνώ. Όχι δεν θέλουμε τώρα να εξεύρουμε κάποιους πόρους φανταστικούς και έτσι να αυξήσουμε το φορολογικό βάρος το οποίο βαρύνει τόσο πολύ φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Και συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε ότι έχουμε στην Ευρώπη πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Δεν το έχουμε λύσει ακόμα. Άρα Άρα να προσέξουμε και την παραγωγή αλλά και την απασχόληση. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε που δεχτήκατε να έρθετε ενώπιόν μας. Δεχτήκατε αυτή την Mission ε, Impossible, την ε, αδύνατη αποστολή, αποστολή που είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Είναι πάρα πολύ συναρπαστικό το εγχείρημα που έχετε μπροστά σας και εμείς θεωρούμε ότι κάποια στιγμή θα πούν όλοι ότι ξέραμε ότι ήταν, δεν ήταν αδύνατο και τα καταφέραμε. Καλό θάρρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, ελάτε και πάλι στην ημέρηση διάταξη η οποία είναι φορτωμένη αφού προηγουμένως καθίστε παρακαλώ. Κύριε Φερνάντς. Κύριε Φερνάντς. Αγνοούμενος ο κύριος Φερνάντς. αναζητείτε ο κύριος Φερνάντες. Κύριε Δεπρέ, θα θέλατε να λάβετε τον λόγο για το σχέδιο εγγράφου κατευθύνσεως σε σχέση με τον προϋπολογισμό 2016, τμήμα 1, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, ήμουν αφηρημένος, αλλά φτάσαμε στο σημείο 10 ήδη. 10 διότι την έκανε ο εισηγητής του σημείο 9 προσωρινά. Α, το κατάλαβα λέει ο κύριος Στέπρε. Α, κύριε εισηγητά, καλώς ήλθατε, σας αναμένω μεν. Όταν πρέπει να μιλήσετε δεν μπορείτε να απουσιάζετε. Κύριε Φερνάντε, λοιπόν, πρώτο για το σημείο 9 και θα ακολουθήσει ο κύριο Δεπρέ, ο έχει το χρόνο να ετοιμαστεί έτσι. Κύριε Φερνάντε, για τι κατευθυντήρε γραμμέ του προπολογισμού 2016, τμήμα 3. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα πορτογαλικά. Η έκθεση αυτή αποτελεί μια ευκαιρία να δώσουμε κατά κάποιο τρόπο μια καλύτερη έμπνευση με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ε, πρόταση της Κομισιόν. Και από αυτή την άποψη μιλάμε για μια πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα σχέδιο προπολογισμού, αλλά έχει εδώ την ευκαιρία να παρουσιάσει ένα σχέδιο προπολογισμού το οποίο θα αντιμετωπίσει και τις προτεραιότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις αιτήσει του Κοινοβουλίου και τι ανησυχίε του Κοινοβουλίου. Αυτές οι κατευθύνσει που δίνουμε στην Κομισιόν ξεκινούν από μια βασική αποδοχή ότι τα προβλήματα που έχουμε με τις πιστώσεις πληρωμών θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και ότι οι δηλώσει του Συμβουλίου επίση θα πρέπει να ακολουθηθούν από πράξεις και όσο μιλάμε για τις ε, πληρωμές είναι απαραίτητο να έχουμε ένα σχέδιο για την εκταμείευση αυτών των πληρωμών. Θα, πάει, θα υπάρξει μια πρώτη διαθεσμική συνάντηση το Μάρτιο και θα πρέπει επιτέλους να λυθεί το πρόβλημα αυτό που έχει να κάνει με το 2015. Ο προϋπολογισμός του 2016 έχει σημεία συμφόρησης που οφείλονται σε αυτά τα προβλήματα που δεν έχουν επιληθεί. Η δομή του προϋπολογισμού μου φαίνεται ότι του εγγράφου μου μάλλον πρέπει να είναι ένα κατά την άποψή μου, ένα έγγραφο απλό με σαφείς επιλογές οι οποίες θα πρέπει να γίνουν κατανοητές. Θα πρέπει να δώσουμε σαφή μηνύματα και στους πολίτες που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά, είναι η προτεραιότητά μας. Θα πρέπει να καταδείξουμε ότι ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει <clears throat> να εξασφαλίσει το ότι θα υπάρξουν επενδύσεις και οι διοικητικές δαπάνες θα πρέπει να είναι περιορισμένες, μόνο το 6%. Το κύριο μήνυμά μας είναι τα 3 ε στα πορτογαλικά. Ε, απασχόληση, επιχειρήσεις, επιχειρηματικό πνεύμα. Η Ευρώπη του 2020 θα πρέπει να στοιχηματίσει στα προσόντα, στην παιδεία και ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες χρειάζονται ένα θετικό επιχειρηματικό κλίμα. Όταν μιλάμε για επιχειρηματικό πνεύμα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για έρευνα, για προγράμματα τα οποία υποστηρίζουμε όπως, και στο, όπως το Horizon 2020 και το COSME. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα το οποίο θα δώσουμε είναι πάρα πολύ σημαντικός και ο ρόλος των διαρθρωτικών πόρων για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Για τα θέματα της απασχόλησης και της απασχόλησης των νέων θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις ανησυχίες και πρέπει να υλοποιήσουμε τα σχετικά προγράμματα. Κυρίως τα προγράμματα κινητικότητας, αλλά η κινητικότητα μπορεί να είναι σημαντική. Η Ευρώπη έχει εκατομμύρια κενές θέσεις κάθε μέρα, όταν από την άλλη πλευρά έχουμε τεράστια ε, ανεργία σε άλλες χώρες μέλη. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο αλλά υπάρχει και μια ευκαιρία. Όταν υπάρχουν άνεργοι και υπάρχουν και θέσεις θα πρέπει να βρούμε τρόπους με τους οποίους θα βοηθήσουμε τους άνεργους να βρουν μια θέση εργασίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι απαραίτητο όμως να σκεφτούμε και τα απαραίτητα προγράμματα για να τονώσουμε την κινητικότητα αυτών που δεν είναι πια νέοι έχουν ξεπεράσει την ηλικία των 30 ετών και θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε προγράμματα και σχέδια τα οποία θα δώσουν δυνατότητα και των πιο μεγάλων σε ηλικία και όχι μονάχα των νέων να έχουν μεγαλύτερη κινητικότητα. Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε και το θέμα της εσωτερικής αλληλεγγύης, τα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τον αγώνα κατά της ένδυας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να είναι ένα σημαντικό στόχος λοιπόν της Ευρώπης 2020. Χρειάζεται επίσης να υπάρχει εσωτερική συνοχή της δράσης των διαχρονικών πόρων και θα πρέπει να ενισχύσουμε την εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ευρώπης με εσωτερική αλληλεγγύη. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε σχέση με την άμεση γειτονιά της, με την Ουκρανία συγκεκριμένα, να αντιμετωπίσει την ανάγκη να δώσει ανθρωπιστική βοήθεια. Κάτι που πάντα έχουμε τονίσει, ότι εμείς είμαστε ο μεγαλύτερος παγκόσμιος δωρητής σε επίπεδο βοήθειας προς τον τρίτο κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν στοιχείο του προπολογισμού η εξωτερική αλληλεγγύη, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από την εσωτερική αλληλεγγύη. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε τη σύνδεση μεταξύ αυτών των δύο να έχουμε μια Ευρώπη η οποία θα είναι ασφαλέστερη με τον τρόπο αυτό. Ο προπολογισμό επίσης το 2016 θα έχει ελπίζω ένα άλλο στοιχείο, το σχέδιο επενδύσεων, την υλοποίηση του σχεδίου Juncker και σε σχέση με το σχέδιο Juncker, αυτά τα οποία λέω στην έκθεσή μου, είναι ότι θα πρέπει να δούμε το σχέδιο Juncker ως ένα συμπληρωματικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος δεν μπορεί ποτέ να αντικαταστήσει πλήρως τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι φανερό ότι ο προϋπολογισμός αυτός έχει να εξασφαλίσει μια δύσκολη ισορροπία. Πρέπει να σεβαστούμε τις υποχρεώσεις μας για να είμαστε αξιόπιστοι. Αν δεν είμαστε αξιόπιστοι δεν μπορούμε πράγματι να δημιουργήσουμε καμία εμπιστοσύνη. Γι' αυτό θέλουμε οι δεσμεύσεις που έχουν ληφθεί ιδίω στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 να υλοποιηθούν. Ο σεβασμός αυτών των υποχρεώσεων σημαίνει ότι όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα, όλα τα ευρωπαϊκά ταμεία, οι σχέσεις εταιρικού χαρακτήρα με τα κράτη-μέλη θα υλοποιηθούν πράγματι πλήρως το 2016 και το 2016 θα μπορέσουν όλα τα προγράμματα που περιέχονται στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο να ξεκινήσουν και να βρουν τη σωστή τους ταχύτητα. Οι δηλώσεις τώρα που ελπίζουμε ότι θα γίνουν σε σχέση με τις πληρωμές από την Κομισιόν θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις πιστώσεις πληρωμών του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Αυτό είναι η ελπίδα μας λοιπόν. Επίσης προσδοκούμε ότι θα υπάρξει το κατάλληλο πλαίσιο και ξέρουμε ότι μέσα στο 2015 θα πρέπει να επιτευχθεί μια συμφωνία για να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο πληρωμών. Όπως έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, είναι απόλυτα απαράδεκτο να υπάρχουν όλα αυτά τα οφειλόμενα ποσά. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο προσπαθούμε να περάσουμε. Φτάσαμε στα 24,7 δισεκατομμύρια απλήρωτων λογαριασμών στο τέλος του 2014. Αυτό είναι κάτι το χωρίς προηγούμενο. Σε σχέση με το δρόμο τώρα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε, ελπίζουμε ότι το 2016 θα λάβει χώρα και η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και θα ακολουθήσει αυτό το πνεύμα ένα πνεύμα τήρησης των υπεσχημένων αναθεώρησης μετά από επισκόπηση των αναγκών και επίσης και της αντιμετώπισης του θέματος των ιδιών πόρων που θα τεθεί το 2017 ήδη. Ελπίζω λοιπόν ότι οι θέσεις μας θα πρέπει να είναι πραγματικές προτεραιότητες, θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα μήνυμα που πρέπει να δώσουμε στους πολίτες μας. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι με αυτά. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει μια απλή διάρθρωση με το στόχο τον οποίο ανέφερα για να μπορέσει η Κομισιόν να λάβει υπόψη αυτά τα οποία έχουμε κάνει σε σχέση με τις γενικές κατευθυντές γραμμές. Είναι απαραίτητο η Κομισιόν λοιπόν να συμπεριλάβει στο λειτουργικό της πρόγραμμα τις ε, αιτήσει και τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις νέες αυτές τις ε, πρωτοβουλίες και τις προτεραιότητές μας και φυσικά είναι απαραίτητο το Συμβούλιο να φέρει σε πέρα στις υποχρεώσεις του ώστε να δημιουργήσει στους πολίτες την εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση και αλληλεγγύη στο εσωτερικό και σε εξωτερικό επίπεδο στην Ευρώπη. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες οι οποίες έχουν συμβάλει στην ε, ορίμανση αυτής της έκθεσης Συνεχίζω φυσικά να αναμένω τις συμβολές των συναδέλφων και στο βαθμό του δυνατού. Ελπίζω ότι οι συνεισφορές των συναδέλφων θα ακολουθήσουν αυτή τη δομή που θέλησα να δώσω στην έκθεση αυτή και που είναι απαραίτητη εν ώψη της συζήτησης που θα χρειαστεί να κάνουμε. Και ακολουθώ αυτά τα οποία λέξαν και στην προηγούμενη μας συνεδρίαση που συζητήσαμε για πρώτη φορά αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντε Υπάρχουν παρατηρήσεις τώρα σχετικά. Η κυρία Γουαρδιά Σαβάλου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς, όπως είπαμε και στην αρχή. είπαμε να κάνουμε διέρεση εργασιών, αλλά τώρα λείπει ο συνάδελφος Γκάγερ και επομένως πρέπει εγώ τώρα να σας πω για το ε, έγγραφο Φερνάντες. Περίπλοκο είναι λέω. Λέμε για καινούριο προπολογισμό, νέες ιδέες και ελπίζω όλοι να είμαστε πιο αναζωογονημένοι τώρα μετά τις τόσο δύσκολες διαπραγματεύσεις που γίνανε. Να μην ξεχνάμε βέβαια τι κουβαλάμε. Τώρα στη συνέχεια της πολιτικής προπολογισμού. Εντάξει, ε, ξεκάθαρο είναι το έγγραφο, είναι καλό, έχει τους στόχους, τις πολιτικές, αυτά που θέλουν να ο κ. Βερνάντες, ε, τις ιδέες του, ε, όλα ξεκάθαρα. Ασχολείται με τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου αρκετά. Βεβαίως και αναδεικνύει τις αξίες και απόψη της πολιτικής του ομάδας. Απασχόληση, επιχείρηση και επιχειρηματικότητα. αλλά δεν λέει τίποτα για την συγκρότηση της οικονομίας, αλλαγές στην οικονομική πολιτική και τόνωση της ζήτησης. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο τώρα κινούμεθα. Άρα θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε τόσο ώστε ο προϋπολογός να μπορέσει να έχει μέλλον. Και λέμε τώρα για τη χρήση του 2016. Αλλά προϋπολογισμός αυτός θα εξαρτηθεί από πολλές μεταβλητές που δεν ξέρουμε ακόμα και πάρα πολλά ερωτηματικά. Θα είναι η πρώτη χρονιά όπως λέει το έγγραφο οπότε και δεν θα υπάρχουν χρήματα τα οποία έχουν προδιατεθεί για την εγγύηση, για την ε, νεότητα αλλά θα έχουμε ένα γενικότερο πλαίσιο για, ε, για τις πιστώσεις υποχρεώσεων αλλά ακόμα δεν γνωρίζουμε τώρα, τώρα που δουλεύουμε δύο χρόνια πριν, ή ένα χρόνο μάλλον πριν, τι θα γίνει με τις ε, επενδύσεις. Ούτε για αυτόν τον υπολογισμό, ούτε για τον επόμενο, καταμίζουν λόγο. Επίσης, παράλληλα, λέμε τι θα γίνει με την αλλαγή του πολιτούς πλαισίου. Επίσης, ταυτόχρονα, έχουμε ένα άλλο μέτωπο, τις πιστώσεις πληρωμών. Οπότε, έχουμε αυτές τις τέσσερις μεταβλητές που θα καθορίσουν κατά πολύ την θέση του Κοινοβουλίου για τον προπολογισμό του 2016. Μιλούμε τώρα για κατευθυντήριες γραμμές. Μιλούμε για ένα έγγραφο που θα ξεκαθαρίσει τη θέση του Κοινοβουλίου και θα δώσει και ένα μήνυμα στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τα λάβει όλα αυτά υπόψη. Αλλά έχουμε πολλές εμφυλίες και όλες αυτές τις μεταβλητές. Χωσέ να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το πρώτο εξάμεινο για να διαμορφώσουμε τον πρόεδρο του 16 οπότε σου εύχομαι καλό κουράγιο στη δουλειά αυτή. Merci, Monsieur Ali. Thank you, Mr. Chair. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υποστηρίζουμε τον εισηγητή στο, δεύτερο, στο θέμα αυτό σε ό,τι αφορά τους γενικότερους, τη γενικότερη γραμμή για τον προϋπολογισμό για το 2016. Είναι καλά δομημένη η έκθεση, οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές και οι επιπρεότητες ε, έχουν σωστή μορφή. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και σε άλλους τομείς έχουν εφαρμοστεί στο έγγραφο αυτό σε αφορά την θέση απασχόληση στη δημιουργία επιχειρήσεων, εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου του Juncker. Αυτό συμπεριλαμβάνεται στο γενικότερο πλαίσιο, που είναι πολύ σημαντικό. Το επενδυτικό σχέδιο του Juncker θα σταματήσει το 2016. Πιστεύω ότι είναι καλά βήματα αυτά. Έχουμε κάποιες τροπολογίες. Όχι πολύ για θέματα ουσίας, πιο πολύ και λεπτομέρειες, τις οποίες συζητήσαμε και με τον εισηγητή. Αλλά γενικά υποστηρίζουμε τον εισηγητή και τις γενικότερες κατευθυντήρες γραμμές για το 2016. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Λίγο ο Δεν ζητάει κανεί άλλο το λόγο. Να σας επισημάνω ότι οι τροπολογίες για την έκθεση του κυρίου Φερνάντε. θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου και θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν στι 26 Φεβρουαρίου και το Μάρτιο θα αποφανθεί η Ολομέλεια για την έκθεση αυτή για τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προεπολογισμό 2016, τμήμα 3. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ντέμπρε. Να περάσουμε μάλλον στην πρώτη ενότητα, σχέδιο προπολογισμού του ε, Κοινοβουλίου για το 2016. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι ότι δεν ήμουνα έτοιμος, αλλά ήθελα προφανώς να αφήσω τον φίλο μας, τον κύριο Φερνάντς, να λάβει το λόγο, γιατί εγώ είμαι απλό εισηγητής για τα άλλα τμήματα και φυσικά ο προπολογισμό της Κομισιόν είναι αυτός που επέχει προτεραιότητα. Αυτή τη στιγμή έχω μονάχα ένα έγγραφο εργασία που θεωρώ ότι είναι αξιοσημείωτο, εν πάση περιπτώσει, τμήμα το οποίο δεν είναι το δικό μου. Αυτό το οποίο εξεπώνησε η γραμματεία της Επιτροπής μας και περιλαμβάνει μερικές πολύ καλά παρουσιασμένες και δομημένες πληροφορίες για την πορεία του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τη στιγμή που ετέθησε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Υπάρχουν συγκριτικοί πίνακες που δείχνουν τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, από το 2011 μέχρι σήμερα, το πώς έχει αυξηθεί ο προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βλέπετε στο έγγραφο επίσης το ιστορικό όλων των προτεραιοτήτων που έχει θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία αυτά χρόνια τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν και αυτό μας δίνει ένα σαφές πλαίσιο για την περαιτέρω εργασία μας. Είναι πολύ ενδιαφέρον λοιπόν αυτό το τμήμα και προσκαλώ όλους τους συναδέλφους να το διαβάσουν μέχρι το σημείο που ερχόμαστε στις πρώτες προκαταρτικές κατευθύνσεις για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2016 και από εκεί πέρα είναι αποκλειστική ευθύνη μου τα γραφόμενα και θα ήθελα να έχω και την άποψη των συναδέλφων μου και των πολιτικών ομάδων. λοιπόν, διευκρινίζω τώρα ότι στο τρέχον στάδιο οι κατευθύνσεις αυτές είναι προκατακτικού χαρακτήρα, βασίζονται σε μία μοναχά συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος θα έλθει ε, συντόμως ενώπιον μας για να υποστηρίξει τις ε, προβλέψεις αυτές για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή μας και έχω κάνει μια σύντομη επαφή με τους σκιώδεις εισηγητές. Έχουμε εντοπίσει μια σειρά από ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία αλλά δεν είχα ακόμα την ευκαιρία να τα συμπεριλάβω στην έκθεσή μου γιατί αυτή η συνάντηση είναι πάρα πολύ πρόσφατη. Λοιπόν, θα παρουσιάσω συνολικά αυτή τη στιγμή το περιεχόμενο των πρώτων κατευθυνσεών που θέλω να σας υποβάλω στη σοφροσύνη των συναδέλφων μου. Η πρώτη προκατακτική λοιπόν κατεύθυνση για τον προϋπολογισμό και εδώ δεν είμαι μεταξύ αυτών <clears throat> που θέλουν να είναι χαλαροί για τα θέματα αυτά. Θέλω οποιαδήποτε αύξηση του προϋπολογισμού να είναι μέσα σε συγκεκριμένα όρια όταν και οι προπολογισμοί των περισσότερων κρατών το, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προπολογισμοί είναι σε πάρα πολύ στενό κορσέ. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ζητείτε να υπάρξει περιστολή της αύξησης του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάτω από το 20% του, της κατηγορίας 5, δηλαδή των διοικητικών δαπανών των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Προτείνω λοιπόν να μην υπερβούμε το 20% των συνολικών διοικητικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άμα κοιτάξετε τον πίνακα που βρίσκεται στο έγγραφο αυτό στη σελίδα 3 βλέπετε ότι είμαστε πολύ κοντά στο 20% το οποίο το είχαμε ξεπεράσει πέρσι ενώ τα άλλα χρόνια ήμασταν στο 19, κάτι τα Προτείνω λοιπόν να μην ξεπεράσουμε καταρχήν το 20% των συνολικών διοικητικών δαπανών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχρόνω προτείνω η αύξηση του προπολογισμού του Κοινοβουλίου του 2016 έναντι του 2015 να μην ξεπεράσει το 2%. Σας λέω γιατί. γιατί. Κοιτάξτε και <clears throat> αυτό βρίσκεται στο πρώτο υπόμνημα της ε, έκθεσης που έχει γίνει από τη γραμματεία της Επιτροπής Προϋπολογισμών μπορείτε να δείτε ότι το 2% σε πραγματικούς όρους είναι κάτι το εφικτό άμα δείτε την αύξηση των κονδυλίων από το 2011 στο 2015. Κάποιοι συναδελφοί μου ίσως μπορεί να μην συμφωνήσουν με αυτό. Πώς έφτασα στο 2%? φυσιολογικά ενσωματώνουμε στον προϋπολογισμό γιατί υπάρχει φυσικά το κόστος του προσωπικού και η Κομισιόν τα έχει προβλέψει αυτά προκύπτει ένα, μια τιμαριθμική αναπροσαρμογή 1,6% για το 2016 αυτό λοιπόν πρέπει να συμπεριληφθεί λόγω της αναπροσαρμογής των ε, αποδοχών του προσωπικού και υπάρχει και μια σειρά προτεραιοτήτων που εγώ αποτιμώ στο 0,4 του προπολογισμού και γι' αυτό <clears throat> προτείνω μια αύξηση, εάν συμφωνείτε βέβαια με τις προτεραιότητες αυτές, 2% για τον προϋπολογισμό του 16 σε σχέση με το 2015. Μία από τις πρώτες προτεραιότητες μου, και έχω ήδη μιλήσει με τον Γενικό Γραμματέα για το θέμα αυτό και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ζητήσει η Επιτροπή μας να το εξηγήσει ο Γενικός Γραμματέας σε μια μεταγενέστερη συνεδρίασή μας. 26 Φεβρουαρίου έχουμε μια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα που θα παρουσιάσει τις προβλέψεις για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως τις προτείνει η Γραμματεία του Κοινοβουλίου. Πρώτη λοιπόν προτεραιότητα είναι η ασφάλεια. Τα πρόσφατα γεγονότα έδειξαν ότι το έγγραφο αυτό σε ό,τι αφορά τον περίγυρό του και την πρόσβασή του έχει σχεδιαστεί σε μια εποχή που δεν ήταν τόσο ισχυρή μέρημνα η ασφάλεια. Επίσης έχουμε πάρει μια απόφαση πολύ σημαντική το 2013 να μην αναλαμβάνει την ασφάλεια μια εξωτερική εταιρεία αλλά να εσωτερικοποιηθεί. Υπάρχει λοιπόν ένα σημαντικό κομμάτι της γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ασχολείται με τα θέματα της ασφαλείας. Όλο και περισσότερο λοιπόν είναι μια δική μας ευθύνη η ασφάλεια αυτή. Θα ήθελα λοιπόν στην παρουσίαση των προβλέψεων για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου να έρθει να μας μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας για τα μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κόστου το οποίο θα πρέπει να καταλογιστεί στον προπολογισμό του 2016 του Κοινοβουλίου. Κάποια από αυτά τα μέτρα πιστεύω ότι είναι απόλυτα δε δικαιολογημένα. Και το κόστος τους επομένως επίσης. Δεύτερη προτεραιότητα και σε πολιτικό επίπεδο ίσως η πιο σημαντική είναι η εξή. Μετά από την θέση σε ισχύ τη Συνδίκη Λισαβόνα, οι ευθύνε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν αυξηθεί πολύ. Είμαστε συνομοθέτε για το σύνολο σχεδόν των αποφάσεων που λαμβάνονται σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Έχουμε λοιπόν μια αυξημένη ευθύνη σε νομοθετικό επίπεδο και μια αυξημένη ευθύνη σε ό,τι αφορά τον πολιτικό έλεγχο γιατί όταν εγκρίνεται νομοθεσία η οποία πρέπει να εφαρμοστεί στη συνέχεια πρέπει να ελέγξουμε τον τρόπο με τον οποίο η Κομισιόν, η οποία είναι αρμόδια, θα φέρει σε πέρα τις ηλυμένες αποφάσεις στις οποίες έχουμε συμβάλει και εμείς. Προτείνω λοιπόν στο πλαίσιο αυτό τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα, να ενισχύσουμε, ξέρω ότι έχει γίνει ήδη σε κάποιο βαθμό, να ενισχύσουμε το προσωπικό των επιτροπών, το, τη γραμματεία των ειδικευμένων επιτροπών, γιατί στο μέλλον θα είναι σημαντική η λειτουργία μας ως νομοθετών, στο μέλλον, αλλά και κυρίως να ενισχύσουμε τον αριθμό των ε, συνεργατών μας που μπορούν πράγματι να ελέγξουν αποτελεσματικά την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων. Γιατί σε ορισμένε περιπτώσει δεν έχουμε γνώση των προγραμμάτων και δεν έχουμε τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε για τον έλεγχο αυτών των αποφάσεων, <clears throat> όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο που είναι θέμα τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, αλλά και των πολιτικών που έχουν ακολουθηθεί. Λοιπόν, ενίσχυση του προσωπικού των κοινοβουλευτικών επιτροπών, ιδίω για τον καλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο και έχουν να κάνουμε το ρόλο μας ως νομοθετών. Παράλληλα, και μέσα στο ίδιο πνεύμα έριξα μια, ένα βλέφαρο στα θέματα των βοηθών, των συνεργατών, των βουλευτών και βρήκα κάποια παράξενα πράγματα τα οποία ίσως θα πρέπει να μας απασχολήσουμε Σε γενικό επίπεδο σας λέω ότι αυτά τα στατιστικά στοιχεία υπάρχουν, δεν τα έβγαλα από το μυαλό μου. Υπάρχουν ήδη σε ένα επίσημο έγγραφο του Κοινοβουλίου. Κατά μέσο όρο κάθε βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 2,33 διαπιστευμένους συνεργάτες και 6,34 τοπικούς συνεργάτες. Βλέπετε λοιπόν τη σχέση μεταξύ των διαπιστευμένων και των τοπικών βοηθών έχει αυτή τη μορφή οι τοπικοί συνεργάτες αναβουλευτές αναβουλευτή πάνε από το 0 ως το 43. Υπάρχει ένας βουλευτής που έχει 43 τοπικούς συνεργάτες. Είμαι στη διάθεσή σας αν θέλετε να σας δώσω ε, τους λόγους για τους οποίους αυτός ο βουλευτής δεν το θεωρεί ότι είναι παράξενο αυτό. Υπάρχουν 16 βουλευτέ που δεν έχουν τοπικούς βουλευτέ, αλλά υπάρχουν και 84 βουλευτέ που έχουν πάνω από 10 τοπικούς συνεργάτες και με μια πρώτη αναζήτηση που έκανα βρήκα αυτούς τους βουλευτές σε, μια, σε ένα πολιτικό σχηματισμό και υπάρχουν επίσης 45 βουλευτές που δεν έχουν κανένα διαπιστευμένο συνεργάτη και έχουν μόνο τοπικούς συνεργάτες. Αλλά όταν πρέπει κανεί να ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο και νομοθετική εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό μου φαίνεται πολύ παράδοξο. Γι' αυτό προτείνω. Και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε αυτό. Και έχω αναφέρει το θέμα αυτό ήδη στον ε, Γενικό Γραμματέα, αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε να γίνεται αυτή η διόγκωση του αριθμού των τοπικών συνεργατών των βουλευτών. Θα πρέπει να υπάρξει κάποιος κανονισμός που να λέει μέχρι πόσους από τους συνεργάτες του Ευρωπαϊκού Κοινο... των Βουλευτών που πληρώνονται με τα λεφτά των φορολογουμένων φυσικά να υπάρχει ένας κανόνας που να λέει ότι πρέπει να υπάρξει και κάποιο όριο για το τι θεωρείται εύλογο για τους ε, διαπιστευμένους ε, συνεργάτες και τους τοπικούς συνεργάτες. Το να έχει κανείς μόνο τοπικούς συνεργάτες, αυτό είναι κατάχρηση των δυνατοτήτων των κοινοβουλευτικών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα θεσμικό ε, δικαίωμα μάλλον δεν έχουμε με τον τρόπο αυτό οι βουλευτές κανένα ουσιαστική, καμιά ουσιαστική δυνατότητα χρησιμοποιώντας τους πόρους των φορολογούμενων να ασκήσουν τη δραστηριότητα των ελεγκτών και των νομοθετών σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Επομένως θα κάνω κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις για το θέμα αυτό. Θα συνεχίσω να, σας, ε, να ακούω τις απόψεις σας και να συζητώ και με τους κοιόδης εισηγητές. Και θα συζητήσω και με την δίκη του Κοινοβουλίου και θα έρθω σε επαφή και με τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος όμως ήδη γνωρίζει ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί κάποια στιγμή αυτό θα περάσει στα ΜΜΕ και θα είμαστε βουτυγμένοι από την κορυφή ως τα νύχια μέσα σε ένα σκάνδαλο και θα είμαστε πάρα πολύ στριμωγμένοι. Κατά πέμπτον, επίσης έχουμε άλλα θέματα, δεν μπορώ να σας τα πω όλα τώρα. Και θα επανέλθουμε γιατί οι συντονιστές και οι οι ηγητές, έχουν υποβάλει τόσα ερωτήματα που θα πρέπει να μαζέψω τα στοιχεία για να απαντήσω, αλλά θέλω να σας πω τέσσερα. Όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είμαστε κάτω από το 20%. Δεύτερον, εξέλιξη του προϋπολογισμού του 2010 για το Κοινοβούλιο, συχνά το 2015 όχι πάνω από 2%. Τρίτον, προτεραιότητε όσον αφορά το προσωπικό του Κοινοβουλίου θα ενισχύσουμε τις γραμματείες των Επιτροπών. Τώρα, για τα νομοθετικά ακόμα δεν έχουμε καταλήξει, αλλά για όλες τις επιτροπές θα πρέπει να δούμε πόσο αποτελεσματική ε, είναι η εκτέλεση. Οπότε θα πρέπει να δούμε αν τα προγράμματα είναι ανάλογα με, με την ε, αποτελεσματικότητα που θέλουμε τόσο η εκτέλεση των προγραμμάτων, αν είναι αποτελεσματική η εκτέλεση του από το Κοινοβούλιο. Ε, Επίση θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει για τη σχέση μεταξύ διαπιστευμένων και τοπικών συνεργατών και επίσης θα πρέπει να δούμε ε, πώς λειτουργεί η Ασφαλτική Βουλή. Ε, έτσι έχει αυτή η διαδικασία, προχωράει, θα κάνει μια έκθεση ε, σε πρώτο στάδιο ο Γενικός Γραμματέας, αλλά επίσης πρέπει να σας διευκρινίσω ότι υπάρχουν εν κάποια σημαντικά ζητήματα όσον αφορά τα κτίρια. Και ο Γενικός Γραμματέας τώρα ασχολείται με το τι γίνεται όσον αφορά τα γραφεία του Κοινοβουλίου, οπότε να έχουμε ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για τα γραφεία του Κοινοβουλίου, ε, τι χρειαζόμαστε παραπάνω. Κάποια κτίρια που έχουν προβλήματα. Γιατί μια φορά δεν υπάρχει ούτε θέρμανση, δηλαδή, δηλαδή είναι αστεία θέματα και το γραφείο του Προέδρου χρειάζεται να υποστεί κάποια ανακαίνιση. Και κάποια άλλη χώρη θα πρέπει βάθρων να αλλάξουν όπως σε κάποιες θέσεις συνεδρίασεις. Θέλουμε περισσότερες καμπίνες μετάφρασης, διερμηνίας κλπ. κλπ. Τώρα, θα μιλήσουμε και για την ε, ασφάλεια όταν θέμα πει τη εκτιμήσεις του. Επίσης χρειάζεται μια έκθεση για το μεσοπρόθεσμο ε, μεσοπρόθεσμη πρόληψη για τα κοινοβούλια. Το Μάρτιο ή στις 6 ε, θα γίνει αυτό ή στις 31, αν θυμάμαι καλά. Αυτές είναι οι πρώτες μου σκέψεις, κύριε Πρόεδρε, και έτσι είμαι στη διάθεση των συναδέλφων, πέραν των όσων έχω ακούσει από τους σκιώδεις εισηγητές. Και να δούμε τι θα γίνει και με τις ε, περικοπές που προβλέπονται σε διάφορες τομείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να δούμε αν έχει κάποιο πρόβλημα ο Γενικός Γραμματέας, τι έχει, έχει κυκλοφορούν ζώα στο γραφείο. Μανκά. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισήγητη για την ε, συνεκτική έκθεση που περιλαμβάνει πάρα πολλές πληροφορίες. Όταν ήμουν εγώ εισηγητής ε, για τον προπολογισμό την προηγούμενη θητεία, το 2010, προετοίμασα λοιπόν και εγώ την έκθεση αυτή και πολύ λυπάμαι που δεν έχει καλυφθεί αυτή η περίοδος. Σύμφωνο όμως με πολλά από τα στοιχεία που περιλαμβάνει η έκθεση, Συμφωνώ ότι ο γενικότερος προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν στο πέμπτο τμήμα 20% και λιγότερο. Καλός κανονισμός αυτός, καλός κανόνας και θα πρέπει να διατηρηθεί λοιπόν. Θα αυξήσουμε στον προπολογισμό του Κοινοβουλίου κατά λιγότερο από 2%. 1,1% υπολογίζεται ο πληθωρισμό στην επόμενη περίοδο στην Ευρωζώνη. Ίσως θα πρέπει να το συνυπολογίσουμε αυτό και ίσως θα πρέπει η αύξηση να είναι παραπάνω από 2%, πολύ παραπάνω. Κάποιο άλλο σχόλιο. Ίσως ε, όπως ε, κάναμε ως τώρα, δεν θα πρέπει να αυξήσουμε τη συνεισφορά τις ε, αμοιβέ των ε, βουλευτών δεδομένε και της ε, τιμαριθμικής προσαρμογής ίσως θα ήταν θετικό μήνυμα ύστερα για τη μείωση του προσωπικού κάθε χρόνο καλούμαστε να μειώσουμε το προσωπικό κατά 1% συνολικά αυτό 5% αυτό ισχύει και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά πιστεύω θα πρέπει να βγάλουμε εκτός της ρύθμισης αυτής τις πολιτικές ομάδες. Έχουμε 6.000 ε, υπαλλήλους. Μπορούμε να μειώσουμε αλλού το προσωπικό. Μπορούμε να αλλάξουμε και να μειώσουμε το προσωπικό κατά 1%. Να βρούμε πιο πολλά μεγάλα αποθεματικά, κάποια άλλα αποθεματικά. Και άλλη μια ιδέα για το πού θα πρέπει να βρούμε τα αποθεματικά αυτά η έκθεσή σας αυτή έχει μεταφραστεί σε μία γλώσσα και οι τροπολογίες έχουν τροπολογία. Θα ψηφίσουμε σε διάφορους, σε κάποιους μήνες, όλες οι τροπολογίες που θα περάσουν θα πρέπει να έχουν μεταφραστεί και στις 23 γλώσσες. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μεταφραστούν αυτές οι τροπολογίες που δεν θα περάσουν σήμερα. Αυτό θα αποτελούσε απόθεμα. Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από εξωτερικούς μεταφραστές να κάνουν τις μεταφράσεις αυτές και ίσως λοιπόν αν δεν μεταφράσουμε και σε 23 γλώσσες ε, μια τροπολογία που δεν θα περάσει μπορούμε να γλιτώσουμε 3 εκατομμύρια ευρώ από πού? Ξέρουμε πολύ καλά ότι ως βουλευτές μπορούμε να θέσουμε ερωτήσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να απαντήσει και η μία απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοστίζει 1.600 ευρώ. Κάποιες φορές τα ερωτήματα αυτά που τίθενται τίθενται μόνο επειδή ο εκάστοτε βουλευτής θέλει να κάνει να υπάρξει κίνηση. Σας υπόσχομαι ότι αν καταργήσουμε αυτές τις περίπτες ερωτήσεις θα γλιτώνουμε 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί τέτοιοι τομείς όπου μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα και τελικά καταλήγουμε σε πολύ ψηλά ποσά. Και κάτι άλλο. Το κατά πόσον ε, το Κοινοβούλιο θα αγοράσει, ...ή θα ενοικιάσει υπηρεσίες, κτίρια και το καθεξής. Όταν νοικιάζαμε τα κτίρια, οι δαπάνε ήταν πιο χαμηλές. Αλλά πρέπει να υπάρχει και κάποιο σχέδιο, κάποιο πρόγραμμα για το τι θα κάνουμε με τα κτίρια αυτά. Ας ρωτήσουμε λοιπόν τον Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μας παρουσιάσει την ε, κατάσταση σε ό,τι αφορά τα ακίνητα του Κοινοβουλίου και τα πόσο να αξίζει τον κόπο να τα αγοράσουμε ή να τα νοικιάζουμε. Αν ε, αποφασίσουμε να αγοράσουμε, στην περίπτωση αυτή σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχουν διάφορα κτίρια τα οποία θα εξετάσουμε, διάφορε συναλλακτικέ. Γιατί κατά το παρελθόν είχαμε μόνο μία επιλογή σε κάποιε περιπτώσει. Σε ό,τι αφορά του πιστοποιημένου και τοπικού ε, βοηθού. Αυτό είναι ανησυχία. Αν ένα ε, βουλευτή έχει 43 βοηθού, αυτό είναι ντροπή. Ντροπή για όλου μα. Θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία προκειμένου να μην ε, βλέπουμε τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Φυσικά και οι τοπικοί βοηθοί παίζουν σημαντικό ρόλο στα κράτη-μέλη και τους χρειαζόμαστε και τους αξιοποιούμε, αλλά να υπάρχει και κάποια λογική. Ξέρετε πολύ καλά, συνάδελφοι, ότι όλα όσα συζητούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολουθούνται και από ένα βιβλίο εγγράφων σε έντυπη μορφή. Αν αυτό αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, γλιτώνουμε πάρα πολύ χαρτί. Γιατί δεν φτάνει λοιπόν τα έγγραφα αυτά να τα έχουμε με email. Και αν κάποιος πραγματικά χρειάζεται την έντυπη μορφή, να το ζητάει ειδικά. Γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις καταλήγει τελικά στα σκουπίδια να τα έχουν αυτά τα έγγραφα μόνο όσοι τα χρειάζονται πραγματικά. Νομίζω ότι έτσι μπορούμε να δείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι ξέρουμε πώς να εξορθολογίζουμε τα έξοδά μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Αγκάρ. Ευχαριστήσω τον κύριο Ντεπρέ. Συγγνώμη, γιατί ο συνάδελφος Γίνος δεν μπορούσε σήμερα να παραστεί πάρα πολύ σωστό το να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Οφειλεί και είναι πρακτική σε πολλά επίπεδα και για το προσωπικό κατ' τη Λισαβόνας. Είναι σωστό το να υπάρξει ενίσχυση του προσωπικού στις επιτροπές αλλά θα χρειαστεί περισσότερα ε, να εμβαθύνουν σε αυτά τα στοιχεία για την ασφάλεια. Κοιτάξτε, να τα σκεφτούμε καλά για την ασφάλεια, γιατί πρέπει να είναι το κοινοβούλιο ανοιχτό στον κόσμο. Γιατί αν είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει μέσα ο κόσμος για την προσωπία και αυτά, αυτό θα μας εμποδίσει. Άρα, για να το ξανασκεφτούμε το όλο θέμα. Και πάλι ευχαριστούμε, όποτε μπορέσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Merci, Madame. Monsieur σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι στις διαβουλεύσεις και στις συζητήσεις της Επιτροπής μας πρέπει να καλούμε τους κοσμήτωρες και τους αντιπρόεδρους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βελτιώσουμε λοιπόν την επικοινωνία και αυτό το ζητώ από τη γραμματεία. Δεύτερο στοιχείο, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια ροή δεδομένων η οποία ενισχύεται ε, κάθε μέρα και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσαρμοστούν τα συστήματα και στο Κοινοβουλίο. Αν δεν θέλουμε χαρτί θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι σε όλα τα μέρη του Κοινοβουλίου οι συνδέσει είναι τόσο ισχυρές που όλοι και στην Ολομέλεια με 2.000 άτομα να έχουν ίντερνετ που να λειτουργεί γιατί σε κάποιες περιπτώσεις βλέπουμε ότι σε σημαντικές ε, συνεδριάσεις ε, δεν έχουμε τελικά σύνδεση. Αυτό μας το έχουν επισημάνει και οι δημοσιογράφοι και για μας φυσικά είναι απαραίτητο αυτό το πράγμα σε ό,τι αφορά και τις επαφές με τους ε, πολίτες. Στο Κοινοβούλιο αυτό οι πιο πολλοί από εμά θέλουν να επανεκλεγούν και γι' αυτό λοιπόν παίζει σημαντικό ρόλο οι προσκεκλημένη, το εκλογικό μας κοινό. Δεν έχουμε όμως ε, κάποιες κατάλληλες αίθουσες συνεδριάσεων. Όταν ε, έχουμε κανεί 6 12 άτομα προσκεκλημένους, πού να πάμε, στο μπαρ. Πουθενά δεν έχει κάποια αίθουσα όπου να μπορεί κανείς ε, να συνεδριάζει αποτελεσματικά με κάποια άτομα και για εκδηλώσεις ε, οι δυνατότητες έχουν περιοριστεί λόγω των μέτρων ασφαλείας. Εγώ θέλω και στο μέλλον να έχουμε τη δυνατότητα να υποδεχόμαστε τους προσκεκλημένους μας και ίσως θα μπορούσαμε να δώσουμε και μια έμφαση στους νέους, ε, στα νέα άτομα για να μπορούν να έχουν καλύτερη επαφή μαζί μας. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε και ένα πλάνο σε ό,τι αφορά το αρνητικό πρόσημο του του Ταμείου Συντάξεων. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μειώσεις και οικονομία και σε ό,τι αφορά τις οδηγούς. Τους έχουμε στη διάθεσή μας από 6 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα. Αλλά να έχουμε η δυνατότητα να έχουμε τις υπηρεσίες των οδηγών 6 έως 8 το απόγευμα και κατά τα άλλα να πρέπει να το ζητάμε επί τούτου αν χρειαζόμαστε πέρα από τις ώρες αυτές. Επίσης, μια άλλη πρόκληση. Θα πρέπει να κάνουμε μείωση 5%. Αν ε, τα επόμενα έτη κάνουμε μείωση 1% ανά έτος, θα δυσκολευτούμε. Θα πρέπει να κοιτάξουμε πού μπορούμε να είμαστε πιο αποδοτικοί. Να κάνουμε επανακατάρτιση, ναι, κατάρτιση κάποιων ατόμων από κλάδους όπου περισσεύουν άτομα σε κλάδους που χρειάζονται άτομα. τα τελευταία 7 χρόνια έχει συμβεί μείωση 4% στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν έχουμε λοιπόν πάρα πολύ μεγάλα περιθώρια για τους πιστοποιημένους βοηθούς. Λυπάμαι πάρα πολύ που κάποιοι συνάδελφοι δεν μπορούν να έχουν πιστοποιημένους βοηθούς γιατί έχουν στις Βρυξέλλες πολύ λίγα λεφτά για να προσλαμβάνουν ε, πιστοποιημένους βοηθούς. Αν ο μέσος όρος είναι έξι βοηθοί, καταλαβαίνω τι γίνεται. Γιατί στις εκλογικές περιφέρειες χρειάζεται να συλλέγουν οι βοηθοί πληροφορίες και έτσι κάποιοι επιλέγουν να δίνουν έμφαση στην πατρίδα τους. Αλλά από την άλλη και στις Βρυξέλλες χρειαζόμαστε άτομα με πολύ καλή εκπαίδευση δεν υπάρχει συνδικάτο, αλλά νομίζω ότι τους όρους πληρωμής θα πρέπει να τους βελτιώσουμε. Θα πρέπει να είναι πιο ελκυστικό να δουλεύει κανείς στις Βρυξέλλες ή, εν πάση περίπτωση, εξίσου ελκυστικό με το να δουλεύει κανείς στην πατρίδα του. Γι' αυτό λοιπόν στο μέλλον θα πρέπει να προσέξουμε προκειμένου εδώ στο Κοινοβούλιο να έχουμε επαρκείς αρκετούς πιστοποιημένους και ικανούς βοηθούς. Ευχαριστώ κύριε Βαλή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε τον κύριο Ντεπρέ. Και όπως και η Αλισάντο με με αυτό το έγγραφο, είναι προκαταρκτικό, οπότε θα συνεργαστούμε ούτως ώστε να μπορέσουμε να το τελειοποιήσουμε τώρα. Έχω κάποιες μικρές αρχικές παρατηρήσεις. Μας λέει εδώ ότι θέλει να υπάρχει μια οροφή για την αύξηση του 2% και σε σχέση και με τον ε, δίκτυ του πληθωρισμού. Τα είπαμε και με τον ε, σκιώδηση ή των σοσιαλιστών. Να δούμε κατά πόσον ε, Κομισιόν θα συμφωνήσει, γιατί έχει, εγώ θα, θα, θα ότι θέλει 1% για τον χρόνο. Δύσκολο να κάνει κανείς προβλέψεις. Είδαμε τι έγινε με την Κεντρική Τράπεζα, τι γίνεται με το τραπεζικό σύστημα. Οπότε θα έχουμε από τη μια μεριά <clears throat> τις δυσκολίες και από την πραγματική οικονομία. Μιλάμε και από πληθωρισμό και στάσιμο πληθωρισμό. Οπότε ίσως εκεί που λέτε για 0,1% θα πρέπει να το αυξήσουν επίσης. Και είπαμε κάτω από τις 100 στο, όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες του του Κοινοβουλίου και επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον έλεγχο για τους τοπικούς ε, συνεργάτες. Ίσως θα πρέπει να έχουμε έναν ε, περιορισμό, μία ποσόστοση και έτσι να αποφύγουμε να υπάρχουν τόσοι πολλοί τοπικοί συνεργάτες. Έτσι κι αλλιώς η εντολή μας είναι εδώ να δουλεύουμε, όχι αλλού. Τώρα τα θέματα της ε, ασφάλειας και τα υπόλοιπα, τα ποντίκια και αυτά, ε, να το, κοιτάξουμε νυφάλια κάποια άλλη στιγμή. Γιατί έχουμε και άλλα θέματα στη διάταξη. Η κυρία Γκρέσλα. Λαμβάνω το λόγο γιατί με τρόμαξε λιγάκι ο κύριος Μάνκα. Εγώ πράγματι δεν θεωρώ να είναι καλό να αποφασίζουν κάποιοι ότι κάποιοι άλλοι δεν χρειάζεται να έχουν πια έγγραφα εργασία. Αυτοί οι οποίοι πρέπει να έρθουν σε μια συνεδρία θα πρέπει να έχουν εγκαίρω τα έγγραφα. Εγώ δεν έχω ίντερνετ στο σπίτι μου. Γιατί οι Γερμανοί χρηματοδοτούν το ίντερνετ άλλων, αλλά όχι το δικό του πολλέ φορέ. Και εγώ ω πρόεδρο τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, μπορώ να σα πω ότι οι συνάδελφοι διαβάζουν όλο και λιγότερο τα ηλεκτρονικά έγγραφα. Δεν μπορεί κανείς να, να κάνει σημειώσεις σε αυτά. Μα για μένα αυτό πολλές φορές είναι το πιο σημαντικό. Όταν διαβάζω ένα έγγραφο, το πιο σημαντικό για μένα είναι να κρατάω σημειώσεις πάνω σε αυτό το έγγραφο. Και θέλω να εστιάσουμε στα κύρια θέματα και όχι στα θέματα τα οποία είναι δευτερεύοντα, όπως είναι η εκτύπωση εγγράφων. Το θέμα είναι το κόστος του προσωπικού γιατί το κόστος του προσωπικού δεν είναι εύκολο να το καλύψει κανείς τόσο εύκολα. Άμα εσείς ε, καταργήσετε πέντε θέσεις, αυτό θα σας δώσει περισσότερο χρήμα από το να καταργήσετε την ε, εκτύπωση των εγγράφων. Γι' αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό το θέμα. Γι' αυτό θέλω να σας ε, προειδοποιήσω για την πρότασή σας αυτή για τα έγγραφα. Ευχαριστώ. Ο σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γενικά, θα ήθελα να υποστηρίξω αυτά που ζητά ο κύριος Τεπρέ στην προσπάθειά του να έχει ένα προϋπολογισμό του 2016 όπως το έχει προδιαγράψει. Θα ήθελα όμως να διαφωνήσω λιγάκι με τον κύριο Μάγκα. Αν κάποιοι από τους συναδέλφους μας έχουν πολύ τοπικό προσωπικό δεν θα πρέπει να νιώθουμε εμείς όλοι αμηχανία για αυτό το γεγονός. Αν υπάρχει ένας κλέφτης στην Εστονία, αυτό δεν κάνει κλέφτες όλους τους Εστονούς. Θα ήθελα λοιπόν να υποστηρίξω αυτό που λέει ο κύριος Δεπρέ, ότι θέλουμε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να ρυθμίσουμε καλύτερα τα θέματα αυτά, αλλά εγώ θα ήθελα <clears throat> να πω ότι αυτό το οποίο έχω διαπιστώσει, ότι η καλύτερη ρύθμιση για να αποκαλύψουμε μια κατάχρηση από ένα πολιτικό είναι να το κάνουμε δημόσιο αυτό το, την κατάχρηση που έχει κάνει ή την απάτη που έχει κάνει. Εάν το προσπαθήσετε να το αντιμετωπίσετε με ένα κανονισμό, θα βρει έναν τρόπο να το παρακάμψει. Αλλά αν το κάνετε δημόσιο, θα τον τιμωρήσουν οι εκλογέ του. Και πιστεύω θα ήταν χρήσιμο να έχουμε τον ε, κύριο Βέλε, ο οποίος Ξέρω ότι ο κύριος Βέλλα έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό και μπορεί να τα αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Ταράμ, ο κύριος Ικεοζάς. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο σύντομα σχόλια. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεπρέ για όλα τα σχόλια που μας έχει προσφέρει και τις προτάσεις που έχει κάνει. Αλλά αφού άκουσα τους συναδέλφους για ορισμένα σημεία κυρίω για τα θέματα ασφάλεια. Πιστεύω ότι για τα θέματα ασφάλειας η ασφάλεια πάει να είναι ασφάλεια όταν μιλάμε για την ασφάλεια. Δεν μπορούμε λοιπόν στα θέματα ασφάλειας να μιλάμε ανοιχτά σε επιτροπές όπως είναι η δική μας. Για τα θέματα αυτά νομίζω ότι πρέπει να γίνονται αυτές οι συζητήσεις και κλεισμένων των θυρών με τα άτομα τα οποία είναι πραγματικά αρμόδια. Και επίσης για τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες υπάρχει διαφορά φάσης μεταξύ των τοπικών και των διαπεπιστευμένων συνεργατών μας εδώ. Αλλά όταν έρθει ο κύριος Βέλε θα ήθελα να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά και υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο μου απασχολεί πάρα πολύ για τους συνεργάτες. Είναι η έλλειψη δυνατοτήτων που δίνουμε σε αυτούς τους νέους βοηθούς. Γιατί κάποιος ο οποίος έχει πανεπιστημιακό τίτλο, εντάξει. Κάποιος όμως ο οποίος δεν έχει δίπλωμα, ακόμα και αν έχει κάνει δύο-τρία χρόνια παραδείγματος χάρη ε, νομική παιδεία, ζητείται ε, εμπειρία τριών χρόνων σε κάποιο άλλο τομέα για να μπορέσει να λειτουργήσει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν δίνουμε δυνατότητες στους νέους τους Ευρωπαίους να εργαστούν εδώ πέρα, τους θέτουμε κάποια πάρα πολύ σφιχτά όρια, τα οποία δεν τους επιτρέπουν να εργαστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια αναθεώρηση του θέματος αυτού και όταν έρθει ο κ. Βέλε θα πρέπει να επανέλθουμε και στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ για αυτή την πλούσια συζήτηση και θα χρειαστούμε και πολύ περισσότερο χρόνο για τα θέματα αυτά. Έχετε να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις κύριε Ντεπρά, έχουμε καταγράψει όλα αυτά που... Έχετε καταγράψει αυτά που έλεγα. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω καταγράψει όλα αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι και τα οποία ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Αλλά νομίζω θα έχουμε και πάλι την ευκαιρία να συζητήσουμε για όλα αυτά τα στοιχεία όταν έρθει ο Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώπιον μας για να κάνει μια έκθεση. Δύο πράγματα. Η ασφάλεια δεν σημαίνει αυτόματα περιορισμό πρόσβασης γιατί το είπαν αυτό διάφοροι συνάδελφοι, δεν πρόκειται για αυτό. Η ασφάλεια μπορεί να σημαίνει κάποια στιγμή ότι αν κάποιος παραβιάσει την ε, είσοδο του κτηρίου δεν θα μπορέσει να προχωρήσει πιο πολύ μέσα στο κτίριο. Η ασφάλεια περιλαμβάνει πολλά στοιχεία και απαντώ στην τελευταία παρέμβαση δεν είναι όλα δημόσια αυτά τα στοιχεία. Δεν πρέπει να είναι όλα δημόσια τα στοιχεία αυτά. Το Πρόεδρο έχει πάρει κάποια απόφαση, έχει ένα αρμόδιο αντιπρόεδρο για τα θέματα ασφαλείας και δική μου πρόταση από προσωπική άποψη αν ακολουθηθεί αυτή η πρόταση θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει και μια κοινοβουλευτική επιτροπή όπως υπάρχει σε κάποια κράτη με βουλευτές οι οποίοι είναι ε, δεσμευμένοι να τηρήσουν το απόλυτο για να συζητούν με τον ε, αρμόδιο αντιπρόεδρο για τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται. Εγώ νομίζω ότι αυτό υπάρχει σε πολλά κοινοβούλια και είναι ένας δημοκρατικός τρόπος για να ελέγχουμε και τα θέματα ασφαλείας. Μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή την παράδοση. Κατά τα άλλα έχω καταγράψει όλες τις προτάσεις και προτού παρουσιάσουν νέες ιδέες εγώ φυσικά θα συνεννοηθώ και με τους σκιώδεις εισηγητές και θα επανέλθω. Ωραία, λέω πρόεδρος. μετά από τις 12.40, 12.45 δεν μπορούν να μείνουν οι διερμηνείς. Πρέπει να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία για έξι εκθέσεις που έχουν να κάνουν με το Ταμείο ε, Παγκοσμιοποίησης. Θέλετε να τις ψηφίσουμε την επόμενη φορά χωρίς συζήτηση ή θέλετε να τις αντιμετωπίσουμε τώρα. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα τις ψηφίσουμε χωρίς συζήτηση της αιτήσεις για προσφυγή στο Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Έχουμε την έκθεση της κυρίας Γκρέσλε, η οποία και αυτή αναβάλλεται. Έχουμε μονάχα να ψηφίσουμε την έκθεση που είχα τιμή να σας παρουσιάσω σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. 49 τροπολογίες έχουμε και προχωρούμε στην ψηφοφορία. Πρώτη παράγραφος. Ο εισηγητής υποστηρίζει. Ψήφι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτη παράγραφος. Τροπολογή μόνο 2. Εδώ έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία. Για το πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ. ηλεκτρονική ψηφοφορία. Le scrutin est ouvert. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά ingredient. Τρίτη παράγραφος, τροπολογία 3. Υπέρ ο συγητής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ingredient. Παράγραφος 4, τροπολογία 4. Κατά ο εισηγητής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 4, τροπολογία 5. Υπέρ ο εισηγητής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παραγραφός 5, τροπολογία 6. Υπέρ ο συγητής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παραγραφός 6, τροπολογία 7, προφορική τροπολογία. Πρόκειται για μια προσθήκη που οδηγεί σε ένα ποσό 24,7 δισεκατομμύριων ευρώ μη εξοφλημένων λογαριασμών που είναι χωρίς προηγούμενο και αφορά το έτος 2014 υπέρο υπέρ ο συγκητής, είναι υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6. προηγείο 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επτά. Τροπολογία 9 υπέρ ο συγητής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οκτώ. Συμβαστική. Α υπέρ ο συγητής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Τοπολογία 10. Α, όχι, όχι, συγγνώμη. Ε, την προ... προηγούμενη. 8. Τροπολογία 11 υπέρ Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτονται. 8. τοπολογία 12 όχι καταπίπτει. Το 13 καταπίπτει, το 12 και το 13 καταπίπτει, πάμε στο 8α. Τροπολογία 14. Υπέρ ο συγκητής, ποιοι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Τροπολογία 15. Εδώ έχουμε μια προφορική τροπολογία. Υπέρ ο Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εννέα. Τροπολογία 16. Υπέρ ο Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 9. Τροπολογία 17. Υπέρ. Σογητής ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχή. Εγκρίνεται. 9. Τροπολογία 18. Υπέρ ο συγητής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9α. Τροπολογία 19. Υπέρ εισηγητής ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Αλφα Τροπολογία προφορική. Υπέρ εισηγητής. Και λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει προσαρμογή ανάλογα όσον αφορά τον ρόλο των δύο σκελών υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ ο συγκητής. Και είναι υπέρ. Κατά. το Τροπολογία 21. Αποχές. Απορρίπτεται. 10. 22. Κατά ο συγκητής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10. Το Τροπολογία 23 υπέρ ο Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. 24. Υπέρ ο συγκριτής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 10. 25. Κατά ο Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10. Τροπολογία 26. Υπέρ ο Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 10. 27. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Τροπολογία 28. Κατά ο συγκητής. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Συμβαστική Β. Υπέρ ο συγκητής. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29. Υπέρος ηγητής Παραγραφός 10. Β. Νέο. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Γ. Τροπολογία 30. Καταπίπτει. 10. Τροπολογία 31. Υπέρος ηγητής Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Τροπολογία 32. Πέρασε Προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 11. Τροπολογία 33. Κατά ο εισηγητής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απόχειας. Απόρριπτο. Τα και 35 πίπνο. Και τώρα έχουμε μια προφορική τροπολογία στο 36. Υπέρ ο Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38 της παραγράφου 11α υπέρ ο Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Καταπίδνε. Απορρίπτεται τέλο πάντων. Ε, 10β υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 11 γάμα, τροπολογία 40, κατά ο εισήτης. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 12. Τροπολογία 41. Υπέρ ο εισήτης. Ποιοι είναι υπέρ. είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12. 42 υπέρ ο συγητής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές Απολύτως. 12. το Τροπολογία 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 Τροπολογία 44 κατά ο συγητής, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 13 τροπολογία 45 καταπίπτει. 13, 46 υπέρ ο συγητής, Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 13, 40, 5. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, το 47 στην τροπολογία 47, όχι εγκρίνεται. Παράγος 13, τροπολογία 48, κατά ο εισηγητής, ποιοι είναι υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτωται. 13α, καταπίπτει. Τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου όπως έχει τροποποιηθεί. Ψηφίζουμε. Ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Πέρα ψηφοφορίας. Πώς είπατε. Εγκρίνεται. Το κείμενο 19-7 με έξι εποχές. Θέλετε το λόγο. Α, δεν λειτουργήσε το μηχάνημά σας. Θέλετε το λόγο. Εκτός μικροφώνου. Α, ε, θα ψηφίζετε αποχή. Άρα θα προσθέσουμε την ψήφα σας στις αποχές. Άρα έχουμε οκτώ αποχές. Τι λέει μου. Έχουμε τις μεταφορές πιστώσεων τώρα. Κυρία σαβάλ. για το τμήμα 3. <clears throat> Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε κάποιες ψηφοφορίες ακόμα. Απλώς ε, έχει να κάνει με τις οργανωτικές αλλαγές λόγω της αλλαγής κομισιών και έχουμε επομέν, την υποστηρίζω επομένως ως εισηγήτρια, λέει η κυρία Γουαρδιά Σαμπάλ. Λοιπόν, ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά, παρακαλώ, ψηφίστε. Προφορία. Μεταφορά. Για το τμήμα 3 η εισηγήτρια του προϋπολογισμού το υποστηρίζει. Πέρας, ψηφίσατε όλοι. Ευχαριστώ. Είσαστε υπέρ, κυρία Γκρέσλε. 23 ψήφοι υπέρ και τρεις αποχές μόνο. Για το... Για τα άλλα τμήματα τώρα, κυρία Χολμάιερ. Αγνοούμενη κυρία Χολμάιερ ο κύριος Φερνάντες. Θα πρότεινα να, το, να τα ψηφίσουμε στην επόμενη συνεδρίαση, να κάνουμε μία αναβολή, λέει ο κύριος Φερνάντες. εφαρμογή του άρθρου 27 του Δημοσιονομικού Κανονισμού χρειάζονται 6 εβδομάδες για την έγκριση. Τι, τι ακριβώς ζητάτε εδώ? Α, η κυρία έχει έρθει όμως. Συμφωνείτε για την αναβολή. Συμφωνώ λέει η κυρία Χόλμαρ. Για τις έξι εβδομάδες, δεν ξέρω αν χρειάζονται, θα μπορούσαμε να το ρυθμίσουμε και πιο γρήγορα. Στις επόμενες συνεδρίασεις της Επιτροπής μας θα ζητήσω συζήτηση του, συνάντηση με τον ε, διαμεσολαβητή, γιατί πρόκειται για μεταφορά ε, ατόμων προσωπικού που θα κοστίσει 90.000. Δεν έχω καταλάβει το τι και πώς και προκειμένου, προκειμένου να είμαι σίγουρη, θα ήθελα να έχω μια συζήτηση πρώτα με την κυρία Βάιλη, γι' αυτό λοιπόν ζητώ πρώτα μια αναβολή σε αυτή τη φάση. Μάλιστα. Τρεμπιέν λέει και ο πρόεδρος. Πολιτική κτηρίων, κυρία Ολμάιερ. Νομίζω ότι το αναβάλουμε. Δεν έχετε καμιά ιδιαίτερη αίτηση. Μα τότε έχουμε τελειώσει. Με την ημερήσια διάταξη. Η επόμενη συνεδρία σήμερα στις 26 Φεβρουαρίου, αν θέλει ο Θεός. Έχετε διάφορα θέματα. Όχι. Δεν υπάρχουν διάφορα. Γεια σας αγαπητοί συνάδελφοι.